Hello everyone. If like... Καλησπέρα. Καθίστε για να ξεκινήσουμε τη συνάντησή μας. Χαίρομαι που βλέπω τόσους πολλούς ε, από σας παρόντες. Θετικό είναι να ξεκινάμε στην Επιτροπή Βιομηχανίας με τόσο μεγάλη συμμετοχή. Αυτό ελπίζω να συμβαίνει σε όλες τις συνεδριάσεις στο Κοινοβούλιο. Ίσως γιατί έχουμε και πολύ ενδιαφέροντα θέματα στην ημερήσια διάταξη για τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο σήμερα. Καθίστε λοιπόν και ταυτόχρονα να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε με την σημερινή ημερήσια διάταξη. Μια μικρή αλλαγή στην ημερήσια διάταξη έχει να κάνει με το ότι δεν θα έχουμε το απόγευμα συζήτηση με τον κύριο Επασάλα και με την κυρία Βέσπινα Σπανού, Γενική Διευθύντρια της DG Connect. Το στόχος της συνάντησης ήταν να εξηγήσουμε πώς ε, πάει η κατάσταση στην Ενίζα. Ο κύριος Λεπασά προτάθηκε ως νέος ε, διευθυντής της. Θα γίνει λοιπόν μια ακρόαση κανονική το Σεπτέμβριο. Με αυτή τη μικρή αλλαγή, δεν ξέρω αν έχετε άλλες ε, αντιρρήσεις, συμφωνείτε έτσι, ωραία. Μπαίνουμε στο επόμενο θέμα της σημερινή συνδέση. Με χαρά καλωσορίζω υπουργού από τη Φιβλαδία, την κυρία Κάτρι Κουλμούνη, υπουργό οικονομικών, υπεύθυνη για θέματα ενέργειας, ε, βιομηχανίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έρευνας, καινοτομίας και του διαστήματος, αλλά και την κυρία Σάνα Μάριν, είναι υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. Υπεύθυνη για την τεχνολογία της πληροφορικής, την ψηφιακή ε, ατζέντα και την κύβερνο ασφάλεια. Σας ευχαριστώ και τις δύο που ήρθατε εδώ για να μιλήσουμε για τις προτεραιότητες της Φιλανδικής Προεδρίας. Συνάδελφοι, να σας θυμίσω ότι υπάρχουν κάποιοι φάκελοι που θέλουν διαπραγμάτευση με την Προεδρία και στους τομείς αρμοδιότητας και των δύο υπουργών. Επίσης προσβλέπουμε στην, στις προτάσεις και στην ακρόαση κατόπιν των νέων επιτρόπων αλλά και το πρόγραμμα εργασίας ε, της Επιτροπής. Είμαι βέβαιο ότι θα έχουμε μια πολύ πυκνή φθινοπορεινή περίοδο. Ξεκινώ με τις φιλανδικές προτεραιότητες από τις δύο υπουργούς. Κυρία Κούλμουνη έχει το λόγο πρώτα. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, με μεγάλη χαρά και τιμή είμαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα. Η Επιτροπή Ήτρε και τα μέλη της έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ε, ε, πολιτικής της Ένωσης στον τομέα μας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Προεδρία βλέπει τον ρόλο του Κοινοβουλίου ως ουσιώδη στην πρόθεση των ε, πολιτικών αυτών προ όφελο των Ευρωπαίων πολιτών. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συναντηθούμε συχνά κατά τη διάρκεια της Προεδρία μας και πέραν αυτής και θα συνεχίσουμε και θα εντατικοποιήσουμε το φιλόδοξο έργο μας μαζί για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Με χαρά έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας τις, τις προτεραιότητες της Φιλανδικής Προεδρίας ε, σήμερα. Έχουμε φιλόδοξους στόχους να κάνουμε την Ένωση ανταγωνιστική μέσα σε ένα ουδέτερο κλιματολογικά ε, περιβάλλον. Η Προεδρία μας ε, θέλει να προχωρήσει για να, να σε μια σωστή και πλήρη μερίσια διάταξη να η του τελευταίου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου είναι ένας από τους καθοριστικούς στόχους της Προεδρίας μας. Σε ό,τι αφορά τους στόχους της Προεδρίας για τα νομοθετικά κείμενα προσβλέπω στο να συζητήσουμε μαζί σας και να ανταλλάξουμε απόψεις για μια σειρά θεμάτων. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, τι χρειάζεται η Ένωση για την βιώσιμη ανάπτυξή της στην Ευρώπη αντιμετωπίζουμε παγκόσμιες προκλήσεις. Πρώτον, την αλλαγή του κλίματος που απαιτεί δράση και παρέμβαση από πλευρά μας. Δεύτερον, τεχνολογικές, οι τεχνολογικές εξελίξεις αλλάζουν πολύ γρήγορα τη ζωή μας μέσω της ψηφιοποίησης, της αυτοματοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης. Τρίτον, η ο παγκόσμιος ανταγωνισμός απαιτεί από την Ένωση να δράσει γρήγορα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε γρήγορα να προχωρήσουμε προς κοινωνικά και ε, περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομία, να ανταποκριθούμε δηλαδή στις παγκόσμιες προκλήσεις της Ένωσης και γι' αυτό πρέπει να θέσουμε μια φιλόδοξη μερίσια διάταξη πολιτικής. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της βιώσιμης ανάπτυξης στο, στο πρόγραμμά μας. Πρέπει να προχωρήσουμε προς μια οικονομία ουδέτερη κλιματικά που να, να, ε, να εξυγχρονίσουμε την ενιαγορά, την ψηφιακή οικονομία με έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία. Να έχουμε ενεργή εμπορική πολιτική σαν εξωτερική διάσταση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, νέα, προσόντα και γνώσεις. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η κοινή δουλειά μας χρειάζεται να μετατρέψει τους στόχους αυτού σε δράση. Η Ένωση πρέπει να προσφέρει απτά αποτελέσματα στους πολίτες και οι πολιτικές μας πρέπει να δημιουργήσουν μια ισχυρή Ευρώπη. Όπως ε, ως Φιλανδική Προεδρία θεωρούμε ότι η υλοποίηση της μελλοντική ατζέντα για την ανάπτυξη θα πρέπει να είναι το κεντρικό στοιχείο της δράσης της νέας πολιτικής. Μέτρα πολιτικής πρέπει να είναι ταυτόχρονα και φιλόδοξα και αποτελεσματικά πρέπει να προσφέρουμε ένα πλαίσιο πολιτικής για τα επόμενα πέντε χρόνια και ελπίζω ότι στο τέλος της χρονιάς ως Συμβούλιο θα έχουμε μια ατζέντα βιώσιμης ανάπτυξης για την Ένωση έτοιμη προς υλοποίηση. Με χαρά θα μιλήσω με λεπτομέρειες για τα πέντε στοιχεία του πλαισίου πολιτικής μας. Ξεκινώ. Σημείο 1. Μετάβαση σε μια κοινωνία ουδέτερη κλιματικά. Η αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος είναι ένα μάστι και ταυτόχρονα μια οικονομική ευκαιρία διότι η καινοτομία θα παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτό για να δώσει νέες ευκαιρίες για την διαμόρφωση βιώσιμης ανάπτυξης. Ταυτόχρονα η μετάβαση σε μια κοινωνία ουδέτερη κλιματικά πρέπει να είναι δίκαιη. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα υπάρχει μια καλύτερη αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων. Ταυτόχρονα οι στόχοι της μείωσης ε, των εκπομπών ε, αερίων διοξιδίου του άνθρωπου στις, ε, όπως συμφωνήθηκε στο Παρίσι πρέπει να είναι και αποτελεσματικές και κοστοαποτελεσματικές. Ταυτόχρονα πρέπει να παρέχουν και να επιτρέπουν οικονομική ανάπτυξη για τις επόμενες δεκαετίες. Ο στόχος της μείωσης είναι μηδενικές εκπομπές το 2050. Αυτό σημαίνει σημαντικές αλλαγές πολιτικές, πολιτικής σε όλους μας μακροπρόθεσμα ιδίω. Αυτό είναι ένα στόχο μα, όπω και άλλα μέρη τη ε, Συμφωνία του Παρισιού πρέπει να προσφέρουμε του χρόνου νέε πολιτικέ και στόχου. Η αλλαγή του κλίματο και η αντιμετώπιση τη είναι μια προτεραιότητα για μα. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με βάση την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και των συναδέλφων όταν το Συμβούλιο υιοθετήσει όπως ελπίζουμε την τελική στρατηγική πριν το τέλος του έτους. Τα κράτη-μέλη και η Επιτροπή θα συνεργαστούν με βάση τους όρους κίνητρα και πλαίσιο που θα εξασφαλίσουν μια ουδέτερη κλιματικά ένωση που θα ευθυγραμμίζεται με τη συμφωνία με τη συμφωνία του, με του Παρισιού θα λάβει ταυτόχρονα υπόψη τις εθνικές θέσεις των κρατών μελών και θα σέβεται τα δικαιώματα των κρατών να αποφασίζουν για το energy mix του καθενός. Η Προεδρία ξεκίνησε να εφαρμόζει αυτές τις ε, καθηγητές γραμμές ε, στα πλαίσια του Συμβουλίου σε μια άτυπη, στην άτυπη συνάντηση στο Υπουργό ανταγωνιστικότητα στο και εξετάσαμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε ανταγωνιστικότητα και μείωση των εκπομπών. Δεύτερο στοιχείο της ατζέντα μας είναι μία πολιτική για την ενιαία αγορά που θα βλέπει μακριά, που είναι ζωτική για την αγωνιστικότητα της Ένωσης να υπάρχει μια λειτουργική ενιαία αγορά με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών, ιδίω των ψηφιακών, που αποτελούν και πρέπει να γίνουν να απόσπαστο τμήμα τη ενιαία αγορά. Η Ένωση έχει σημαντικό ρόλο στο να συμβάλλει σε ένα ευνοϊκό κλίμα για τι επιχειρήσει και ταυτόχρονα οι επενδύσεις των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων παίζουν καθοριστικό ρόλο για τη μετάβασή μας σε μια ουδέτερη κλιματικά οικονομία. Τρίτον, δύο λόγια για την σύγχρονη βιομηχανική πολιτική μας και την ψηφιακή οικονομία με έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία. Πρέπει να θέσουμε τους στόχους της Ευρώπης, να γίνουμε δηλαδή ένας ηγέτης, ένας πρωτοπόρος στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία με την τεχνητή νοημοσύνη και τις πλατφόρμες που είναι βασικοί παράγοντες για την επιτυχία της ευρωπαϊκής αγοράς. Η Ένωση πρέπει να διαμορφώσει δράσεις πολιτικές για την πρόσβαση δεδομένων, την χρήση δεδομένων, την νέα χρήση δεδομένων και την διαλειτουργικότητα και εμπιστοσύνη των δεδομένων. Οι αρχές πολιτικής δεδομένων είναι κάτι που απαιτείται διότι οι κοινωνίες μας γίνονται όλο και περισσότερο δικτυωμένες και ψηφιοποιημένες ταυτόχρονα. Επιπλέον, Θέλω να βελτιώσουμε την τεχνική νοημοσύνη. Πολλή λόγος γίνεται για την τεχνική νοημοσύνη, θα αλλάξει τη ζωή μας όντως, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να βελτιώσει την ε, ζωή μας και να, γι' αυτό πρέπει να δούμε τις προκλήσεις που έχουμε ως Ευρωπαίοι πολίτες. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να βοηθήσει τη διαμόρφωση βροντολογικών κανόνων και εμπιστοσύνη στα πλαίσια της τεχνητή νοημοσύνη, με έναν ευρωπαϊκό δρόμο για την ψηφιακή οικονομία που θα γίνει ανταγωνιστικό μα πλονέκτημα. Αυτό όμω απαιτεί μεγάλη έρευνα και ανάπτυξη που ελπίζω να πετύχουμε. Οι καθηγητήρε γραμμέ για το, τη διοντολογία της τεχνικής νοημοσύνης είναι βασικό στοιχείο στην πολιτική μα Τέταρτον, προσόντα. Βασικό στοιχείο της ανάπτυξης σε μια ψηφιακή εποχή η ανάπτυξη, η συνεχής ανάπτυξη των προσόντων είναι κάτι απαραίτητο. Η συνεχής μάθηση θα είναι στο κέντρο της ε, μάθησης στο μέλλον. Ε, με την, πιστεύω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα βιομηχανία, νέους χώρους βιομηχανίας. Πέμπτον, η εμπορική πολιτική, καθοριστικό ρόλο για την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης στα, προς τα έξω, που πρέπει να συνοδεύεται από φιλόδοξη εμπορική πολιτική με πολυμέρεια και με βάση τους κανόνες. Η Ένωση πρέπει να παραμείνει ισχυρός δρόν στην παγκόσμια σκηνή. Η άτυπη συνάντηση Υπουργών Υπεύθυνων για την Αγωνιστικότητα στο Ελσίνκι στις 4 και 5 Ιουλίου πριν από δύο εβδομάδες έδωσε την πρώτη ευκαιρία για τους υπουργούς μας να μοιραστούν μεταξύ του ιδέε για τι προτεραιότητε του προγράμματος εργασία τη επόμενη επιτροπή. Οι Υπουργοί καλωσόρισαν τη συνολική προσέγγιση για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Προβλέπουμε στην συνέχιση τη δουλειά για μια βιώσιμη ε, ανάπτυξη και τη σχετική μερίσια διάταξη και στι συναντήσει του Συμβουλίου τον Νοέμβριο. Δύο λόγια για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, και τον προπολογισμό της Ένωσης. Η ολοκλήρωση του επόμενου Πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου είναι ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς στόχους της Προεδρίας μας. Τον ε, Οκτώβριο θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε τις ε, σχετικές διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο και θα ε, προσπαθήσουμε να καλύψουμε όλα, να βρούμε μια σωστή ισορροπία και μια εκτεταμένη συνένεση στον τομέα που ενδιαφέρει την Επιτροπή σας. Επίσης πιστεύουμε ότι θα πρέπει να μπορέσουμε ο προπολογισμό να παράσχει υλοποιήσει στι πολιτικές προτεραιότητες. τα μελλοντικά προγράμματα λοιπόν του ΠΔΤ θα πρέπει να καλύπτουν και να υλοποιούν και τους στόχους για το κλίμα. Άρα το 25% των δαπανών του προπολογισμού της Ένωσης θα πρέπει να ασχολείται με τις δραστηριότητε αυτές. Ταυτόχρονα πρέπει να προωθήσουμε, να προωθήσουμε την έρευνα και την ανάπτυξη, το Horizon Europe, που είναι ένα εργαλείο ουσιαστικό για την προώθηση της έρευνας. Ταυτόχρονα το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα συμβάλλει στην κοινοτομία παρέχοντας βασικές υπηρεσίες και δεδομένα, αλλά και λύσεις για την αντιμετώπιση του κλίματος. Είμαστε μια επιστημονική πηγή γνώσης και πρέπει να επιδιώξουμε την αριστεία για οικονομική επιτυχία σε, που απαιτεί διατομιακή συνεργασία. Κλείνοντας, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα έλεγα το εξή. Χρειαζόμαστε οικονομική ανάπτυξη που πρέπει να είναι βιώσιμη περιβαλλοντικά και κοινωνικά χρειάζομαστε μια, ναι, ένα νέο σχεδιασμό επιχειρησιακής δράσης που θα βοηθά την κοινωνία. Ας το κάνουμε όλοι μαζί, είμαι έτοιμοι να συνεργαστούμε. Πρέπει να ενισχύσουμε μια ένωση περιβαλλοντικά και κοινωνικά συμπεριλαμβάνοντα όλους προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών ο ρόλο σα ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ω Επιτροπή Ήτρε είναι καθοριστική για την επίτευξη των στόχων αυτών. Ευχαριστώ για την προσοχή σα και προσβλέπω στι συζητήσει μα. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Κουλμούνη. Θα παρακαλούσα τώρα την κυρία Μαρίν να μας παρουσιάσει τους δικούς της τομείς αρμοδιότητας σας. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σήμερα για να συζητήσω μαζί σας τις προτεραιότητες της Φιλανδικής Προεδρίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ψηφιακή επανάσταση που αντιμετωπίζουμε μας προσφέρει και πολλές δυνατότητες. Ταυτόχρονα ε, αμφισβητεί η παραδοσιακά μοντέλα και μας αναγκάζει να προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας σωστός δρόμο για να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να ενώσει την ενιαία αγορά ε, καθώς και την πολιτική ε, για τη βιομηχανία, την καινοτομία και ε, τον ψηφιακό τομέα. Η ψηφιοποίηση αποτελεί και απαραίτητο κομμάτι της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν. Είναι απαραίτητο να βρεθεί ισορροπία ανάμεσα στην προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως είναι το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την ελευθερία του λόγου και τις τάσεις ε, στην ψηφιακή ανάπτυξη. Επίσης, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η ψηφιοποίηση μπορεί να αυξήσει την ανθρώπινη ευημερία. Γι' αυτό η οικοδόμηση εμπιστοσύνη ε, θα πρέπει να είναι ο οδηγός μας ε, στην ψηφιοποίηση, διότι οι άνθρωποι θα μπορέσουν ε, να δρέψουν τα πλεονεκτήματα της ψηφιοποίηση μόνο αν μπορούν να εμπιστευτούν την τεχνολογία ψηφιακές ε, πολιτικές ε, όσον αφορά την χρήση δεδομένων ε, και την ανάπτυξη δικτύων, τον ιδιωτικό βίο και τις ευρυζωνικές συνδέσεις, αυτά θα αποτελέσουν το επίκεντρο των εργασιών μας. Πρέπει να μεταβούμε σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών και τελικά σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών από την ε, οικονομία ε, ορυκτών καυσίνων που έχουμε αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να ασχοληθούμε και με την αυτοματοποίηση και με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους μας ως προς το κλίμα ε, και να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και γι' αυτό θέλουμε ευφύς συνδέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη. Τα δεδομένα είναι η πρώτη ύλη για την ε, ψηφιακή ανάπτυξη και για να έχουμε μια οικονομία δεδομένων θα πρέπει να έχουμε ανθρωποκεντρικές πολιτικές. Θα πρέπει δηλαδή να είναι εύκολο για τους πολίτες να διαχειρίζονται τη χρήση των δεδομένων τους. Άλλε σημαντικέ πτυχέ ε, της πολιτικής για τα δεδομένα είναι η διαλειτουργικότητα, η δίκαιη πρόσβαση και η ποιότητα των δεδομένων. Πιστεύω ότι το κλειδί για μια επικοδομητική συνεργασία είναι το να έχουμε κοινό όραμα. Και όσον αφορά την πολιτική για τα δεδομένα, ε, ο ανθρωπογενικός χαρακτήρα θα μπορούσε να είναι ε, κοινό τόπο για όλου. Άλλωστε, οι εργασίε μα θα πρέπει να καλύπτουν τι ανάγκε των πολιτών. Θέλουμε λοιπόν οριζόντια προσέγγιση και να ασχοληθούμε με ζητήματα όπου πρέπει να γίνουν ε, ακόμα εργασίες, λαμβάνοντας υπόψη ε, τον διατομιακό ρόλο της οικονομίας ε, των δεδομένων. Στόχο τη Φιλανδία είναι να ξεκινήσουμε συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τι αρχέ τη ψηφιακή οικονομία. Τέτοιε βασικέ αρχέ ω προ τα δεδομένα θα δημιουργήσουν ένα νέο πρότυπο για την ε, οικονομία δεδομένων. Η Φιλανδική Προεδρία ε, έχει δεσμευτεί να συνεχίσει τις εργασίες ε, πάνω σε σημαντικά εκρεμή ζητήματα. Μία από τις προτεραιότητές μας είναι η ανάπτυξη υποδομών πέμπτης γενιάς και σχετικών υπηρεσιών. Στόχος μας είναι λοιπόν να ολοκληρώσουμε τον κανονισμό για ε, την ε, διευκόνηση της Ευρώπη της Ευρώπης αν υπάρξει συμφωνία όσον αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο το φθινόπωρο. Όσον αφορά το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη, επίσης είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε τις εργασίες, ε, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια τις ε, διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα συνεχίσουμε τις εργασίες όσον αφορά την πρόταση για την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα και θέλουμε να διασφαλίσουμε νομοθεσία ασφαλείας συνεχίσουμε επίση τι εργασίε πάνω στο Κέντρο Ικανοτήτων για την Ευρωπαϊκή Κυβερνοασφάλεια και ε, ελπίζουμε να επιστρέψουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με εσά στο θέμα αυτό και να καταλήξουμε σε μια κοινή λύση. Όσον αφορά την ανάπτυξη δικτύου 5G στην Ευρώπη, θα πρέπει να σκεφτούμε την ασφάλεια των δικτύων με βάση τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά το Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας, Θέλουμε να προχωρήσουμε περισσότερο εις βάθος στη συζήτηση, ιδιαίτερα όσον αφορά την πολιτική τα δεδομένα και τα δίκτυα 5G. Ε, το Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί υπό Φιλανδική Προεδρία στις 3 ε, Δεκεμβρίου. Επίσης ε, θα οργανώσουμε διάφορες εκδηλώσεις και θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία να σας καλέσω να συμμετάσχετε στη συζήτηση κατά τη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων. Η Φιλανδική Προεδρία θα οργανώσει μια διάσκεψη υψηλού επίπεδου για την οικονομία δεδομένων. Ε, επίσης, ε, θα έχουμε τις ε, ημέρες ψηφιακής μεταφοράς για την ψηφιοποίηση των μεταφορών. Θα εξετάσουμε επίσης συστήματα ψηφιακής διακυβέρνησης. Κυρία Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, θα ήθελα να ακούσω τις προσδοκίες σας και τις ανησυχίες σας και θα κάνω ό,τι μπορώ για να τις λάβω υπόψη ε, κατά τη διάρκεια των εργασιών μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Well, thank you. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ και τις δύο για τις παρουσιάσεις. Εκτιμούμε όλα όσα μας είπατε. Νομίζω ότι είναι τμήμα και της κοινή συνεννόησης και των προτεραιοτήτων που έχουμε καθορίσει για την ευρωπαϊκή πολιτική στο τομέα ε, στους τομείς μάλλον που ενδιαφέρουν την Επιτροπή μας. Πριν ξεκινήσει η συζήτηση με τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και τους συντονιστές, Ω εισηγήτρια για τον προπολογισμό για το 2020, πρέπει να σας πω ότι δεν εκτιμούμε το γεγονός ότι το Συμβούλιο έκανε περικοπές στις δεσμεύσει υποχρεώσεων για τον τίτλο 1α που είναι ε, της δικής μας της εντολής. Έχουμε 747,4 εκατομμύρια ευρώ και πρέπει να σας πω ότι επειδή το 2020 είναι η τελευταία χρονιά πριν από την έναρξη του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, που κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσει ε, με λιγότερα προγράμματα το 2021. Θεωρούμε ότι είναι ζωτική σημασία στο γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του 2020 θα πρέπει να χρησιμοποιήσει πλήρως το διαθέσιμο ανώτατο όριο του τίτλου 1α. Αυτό είναι το μήνυμά μας, ε, το οποίο θα ήθελα να δώσω εξ ονόματος όλης της Επιτροπής. Θα θέλαμε, ε, αν Μπορείτε να κάνετε ό,τι γίνεται στη διάρκεια της συνδιαλλαγής ε, για τον προπολογισμό αργότερα εντό του έτους, ώστε ε, το τελικό ποσό να είναι φιλόδοξο για να δώσουμε ε, κονδύλια για έρευνα και κοινοτομία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πέραν αυτού, Νομίζω ότι τώρα μπορούμε πλέον να ανοίξουμε το, τη συζήτηση με ερωτήσεις και παρεμβάσεις από τις πολιτικές ομάδες. Θα έχουμε ένα πρώτο γύρο σχολείων από τους συντονιστές ή τους εκπροσώπους των συντονιστών και θα ήθελα να ε, μιλήσετε το πολύ τρία λεπτά ο καθένας και ξεκινάμε με τις πολιτικές ομάδες, με τη σειρά, όπως ε, προβλέπεται αναπολιτική ομάδα, η κυρία Φιένα Βίρκυνεν από το ΕΛΚΙ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, καλώς ορίσατε ε, Υπουργή Κολμούνη και Μαρίν και σας ευχαριστούμε που μας παρουσιάσατε τις φιλανδικές προτεραιότητες της Προεδρίας. Τρεις ερωτήσεις έχω. Πρώτον, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Προφανώ ε, θα είναι και μία από τι πιο σημαντικέ αποφάσει οι οποίε θα ληφθούν ε, τις επόμενες μήνες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Βιομηχανία πιέζει για μία αλλαγή προ μελλοντικέ επενδύσει. Ε, το Connecting Europe Facility, η ψηφιακή Ευρώπη, τον ορίζοντα 2020, τον ορίζοντα Ευρώπη. θα θέλαμε να ξέρουμε αν θα διατηρήσετε εσεί αυτό το επίπεδο φιλοδοξία και να εξασφαλίσετε κατάλληλη χρηματοδότηση. Όπω ξέρετε η Φιλανδία ήταν μία από τι χώρε, οι οποίε ήταν διατεθειμένη να κόψει ε, ε, τα κονδύλια του Connecting Europe Facility. Ε, θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον είστε διατεθειμένοι να επενδύσετε περισσότερο σε αυτού του τομεί, οι οποίοι είναι ζωτική σημασία για το μέλλον μα, όπω για παράδειγμα υποδομέ, έρευνα, το Connecting Europe Facility, το πρόγραμμα για την ψηφιακή Ευρώπη, το Ορίζοντα Ευρώπη, ή αν σκοπεύετε να προχωρήσετε σε περικοπές. Μετά, για τη βιομηχανία. Αναφερθήκατε σε βιώσιμη ανάπτυξη και ο Φιλανδό Πρωθυπουργό επίση είπε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Φιλανδική Προεδρία θέλει να εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών. Υπουργέ Κολμούνη, εσεί αναφερθήκατε σε αυτή την πολιτική ε, και το τι καλύπτει, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να γνωρίζουμε τι συγκεκριμένε δράσει πρέπει να αναλάβει η Προεδρία για να επιτευχθεί αυτό ο στόχο. Ποια είναι λοιπόν τα πιο σημαντικά στοιχεία τα οποία θα προωθήσετε τώρα τους επόμενους μήνες προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί στο μέλλον. Και όσον αφορά το κλίμα, η Φιλανδική Προεδρία ανακοίνωσε ότι και η Φιλανδία υποστηρίζει τη μείωση ε, Ε, από το φθινόπερο, αλλά βέβαια θα πρέπει να εξασφαλίζεται και ο ανταγωνισμό ε, κατά τη μετάβαση. Γνωρίζουμε όμω ότι από πλευρά Συμβουλίου δεν έχουν δεσμευτεί όλα τα κράτη-μέλη. Πώ σκοπεύει λοιπόν η Φιλανδική Προεδρία να πείσει όλα τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν σε αυτή τη δέσμευση πριν από την COP25 το Δεκέμβριο φέτο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βίρκουνεν. Η κυρία Τόγια τώρα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, να χαιρετήσω και εγώ με τη σειρά μου τις υπουργούς που εκπροσωπούν εδώ τη Φιλανδική Προεδρία με ευχή για ε, πολύ καλή και καρποφόρα δουλειά. Ε, εκτίμησα πολύ κάποια πράγματα και κάποιε δηλώσει προθέσεων, το γενικότερο πλαίσιο, αλλά θα ήθελα όλα αυτά τα ωραία λόγια κάποια στιγμή να υλοποιηθούν. Επομένω, οι ερωτήσει μου θα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένε, γιατί θα ήθελα να ρωτήσω πώ οι αρχέ αυτέ θα γίνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο σε νομοθετικό επίπεδο ε, και ε, τι θα γίνει στο επόμενο εξάμεινο, το οποίο χαρακτηρίζεται και λίγο από συγκεκριμένα θεσμικά ραντεβού, πολύ συγκεκριμένα. Πρώτη ερώτηση. Αναφερθήκατε σε βιομηχανική πολιτική. Ε, κατά την άποψή μου αφιερώσατε ελάχιστο χώρο στο έγγραφο το οποίο μας υποβάλλατε, αλλά ούτως ή άλλως αναφερθήκατε στη βιομηχανική πολιτική και γνωρίζετε ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου έχουν προβλέψει και μία ανακοίνωση για τη βιομηχανική πολιτική. Ε, ακούγεται όμως ότι τελικά ίσως δεν γίνει. Εσείς τι δέσμευση θα αναλύετε ε, ώστε η Ευρώπη να προτείνει πολύ συγκεκριμένε γραμμές. Τα τελευταία χρόνια τη νιώσαμε την έλλειψη μιας βιομηχανικής πολιτικής θα το πούμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έγινε πολιτική για την καινοτομία, για την ενέργεια, για τα ψηφιακά θέματα, αλλά δεν ε, ε στοχεύσαμε σε, αυτά τα βασικά, σε αυτό το βασικό ιστό για την ήπειρό μα. Ε, τι σκοπεύετε να κάνετε αυτά και κυρίω για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Τώρα, έρευνα. Το Κοινοβούλιο έχει προβλέψει 120 δις ε, πρικοδότηση. Πολύ ε, φιλόδοξη. Αν περάσουμε από την έρευνα και την επιστήμη και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων σε βιομηχανικά αποτελέσματα, τι δέσμευση θα αναλάβετε εσείς ώστε πραγματικά να είναι φιλόδοξος ο προπολογισμό στα θέματα αυτά. Ε, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πολλές προεδρίες είδαμε στην προετοιμασία των ε, ετών προϋπολογισμών τελικά να υποκύπτουν στο τέλος, να κάνουν ένα μικρό δωράκι σε κάθε χώρα και τελικά να μην κάνουν ένα δώρο στην ανάπτυξη και τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελευταία ερώτηση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Αναφερθήκατε ακροθυγώς ε, για τον κανονισμό για τα θέματα και τις αρμοδιότητες. Θα ήθελα πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Το θέμα αυτό έχει μπλοκάρει από το Μάρτιο, δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις γιατί υπάρχει αντίθεση για τις αρμοδιότητες του κέντρου και τη χρηματοδότηση και τις λειτουργίες του. Τώρα, υπήρχε η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας. Το θέμα είναι πώς θα επιληθεί το θέμα, διότι αναφερόμαστε στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, που είναι μόνιμη απειλή, αν δεν υπάρξει κάποια παρέμβαση, αλλά εδώ και μήνες έχει σταματήσει το θέμα, γιατί δεν ξέρουμε ποιος χρηματοδοτεί τι και τι θα κάνει το κέντρο. Είναι μεγάλη αδυναμία της Ευρώπης σε σχέση με τις φιλοδοξίες σας. Δεν είναι δευτερεύον αυτό το θέμα, διότι αν δεν υπάρξει αυτό το κέντρο αρμοδιότητας, θα πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε για τη σημασία της στον κυβερνοχώρο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Τόγια. Από το Renew Europe η κυρία Λαμπάγεβα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Υπουργοί Κουλμούνη και Μάριαν, σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μας και ευχαριστώ και για τις εναρκτήριες παρεμβάσεις Πρέπει να πω ότι ε, είναι εξαιρετικός τρόπος να ξεκινούμε με κυρίες στο Προεδρείο, διότι όταν συζητούμε θέματα όπως ενέργεια, βιομηχανία, τηλεπικοινωνίε, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ε, διάστημα και έρευνα, συνήθως ε, έχουμε άνδρες περισσότερους. Και επειδή η ομάδα μου θέλει να ανανεώσει την Ευρώπη, θεωρώ ότι αποτελεί εξαιρετική αρχή και σας ευχαριστώ πολύ. Η Φιλανδική Προεδρία ε, θεωρεί ότι η βασική της προτεραιότητα είναι η βιώσιμη Ευρώπη, ε, ένα βιώσιμο μέλλον. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα μου. Εγώ κυρίως ε, ασχολούμαι με τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη που θα οδηγήσει, που θα, στις οποίες θα μας οδηγήσει μια βιώσιμη Ευρώπη. Τώρα, τι σχέδιο έχετε για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, δεδομένου ότι αποτελείται κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οικογενειακές επιχειρήσεις, αλλά από την άλλη περιλαμβάνει και πολύ σημαντικούς τομείς, όπως η άμυνα. Ε, γνωρίζετε ότι το Συμβούλιο ενέκρινε κάποια συμπεράσματα προσφάτω επ' αυτού. Η Φιλανδική Προεδρία θα πιέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όντω να μα βοηθήσει να έχουμε αποτελέσματα για τα θέματα αυτά. Για να μπορέσουν να εργαστούν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο οι μικρομεσαίε επιχειρήσει, πρέπει να έχουμε κατάλληλε προποθέσει. Τα διάφορα προγράμματα για τα οποία είναι αρμόδια η Επιτροπή πρέπει να έχουν καταρχά επαρκή προπολογισμό, να σύντομα και να υπάρχει και πλήρη υποστήριξη από τα κράτη-μέλη. Πιο συγκεκριμένα, θεωρώ ότι η Φιλανδική Επιροεδρία θα πρέπει να εργαστεί σκληρά ώστε να εξασφαλίσει το πρόγραμμα για την ψηφιακή Ευρώπη θα λειτουργήσει, ε, διότι δεν έχει προσελκύσει μεγάλη προσοχή εκτό των Βρυξελών, αλλά έχει τεράστιε δυνατότητε. 9,2 δι ευρώ δεν είναι μεγάλο ποσό και το ποσό δεν θα πρέπει να θεωρείται κόστος αλλά επένδυση σε ζωτικούς τομείς της τεχνολογίας και της ανάπτυξης. Ε, μιλώντας για επενδύσει, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονό ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόρο απέχουμε από το στόχο τη επένδυση του 3% του ΑΕΠ στην έρευνα και στην καινοτομία. Για παράδειγμα, σε τηλεπικοινωνίες, στο 5G, στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο κλπ. Χρειαζόμαστε να γίνουν πολύ περισσότερα. Η δεύτερη ερώτησή μου είναι εάν η Φιλονδική Προεδρία θα εστιάσει σε αυτά τα θέματα και στο στόχο του 3% εντό του θεματολογίου του Συμβουλίου. Τέλο, ελπίζω ότι πραγματικά η Φιλανδία θα έχει ευκαιρία να κάνει διαπραγμάτευση για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο και θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να εξασφαλίσετε ότι όλα τα προγράμματα ε, τα οποία αφορούν την Επιτροπή Ήτρα θα ε, είναι προτεραιότητα για του Υπουργού Οικονομικών ώστε να ξεκινήσουμε σοβαρέ ε, συζητήσει για τον μακροπρόθεσμο προπολογισμό τη Ένωση. Σα ευχαριστώ για την περιουσία σα, σα εύχομαι ό,τι καλύτερο και καρποφόρε εργασίε για το επόμενο εξάμεινο και φυσικά είμαστε στη διάθεσή σας για συνεργασία. Ευχαριστώ. Ο κ. Λίνης από τους Πράσινους. Κυρίες Υπουργοί, χαίρομαι που σας βλέπω εδώ για να παρουσιάσετε το πρόγραμμα της ε, Φιλανδικής Προεδρίας. Φιλόδοξο πρόγραμμα, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δράση για το κλίμα και ταυτόχρονα την έμβαση για την έρευνα, την έμβαση για την έρευνα που είναι πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας. στην Επιτροπή μας. Έχουμε και σημαντική πλέον παροχή, η παρουσία γυναικών υπουργών και αυτό είναι ένα καλό βήμα για τη Φιλανδία. Ελπίζω να γίνει και για την Ευρώπη. Μια σειρά ερωτήσεων για το κλίμα και την αρχή της καινοτομίας στην πολιτική της Ένωσης. Η Προεδρία στο πρόγραμμά της θέλει να θέσει το 2050 ως στόχο για μια ουδέτερη κλιματικά Ευρώπη με μείωση κατά 50%, 55% μείωση των εκπομπών σε σχέση με το 2030. Εμείς δίνουμε μεγάλη έμφαση στην αλλαγή της προσέγγισης της ε, έρευνας και ένα βιώσιμο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Η Επιτροπή στις συστάσεις της για, τη, τις πολιτικές κλίμα, κλίμα, για το κλίμα των κρατών μελών τόνισε πολλές ελλείψεις όχι μόνο σε ό,τι αφορά τους στόχους για το κλίμα και τα ανανεώσιμα, αλλά κυρίως την αποτελεσματικότητα της ενέργειας όπως προκύπτει από τα εθνικά προγράμματα αντιμετώπισης του κλίματος. Λίγα μόνο κράτη-μέλη έχουν ε, συγκεκριμένους στόχους, οπότε η συνολική ε, αξιολόγηση δείχνει ότι υπάρχει μια απόκληση κατά 6% σε σχέση με τους στόχους της Ένωσης, μείωση δηλαδή 26% στην Ένωση εκτός από το 32,5% όπως ελάχιστος, ελάχιστο στόχο. Αυτό σημαίνει ότι πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα. Πώς η Προεδρία λοιπόν θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα, τι θα κάνει για να εξασφαλίσει ότι οι εθνικές συνεισφορές αυξάνονται για να καλύψουν την τρύπα που υπάρχει. Η άλλη ερώτησή μου αφορά στην αρχή της καινοτομίας που συζητήσαμε στο πλαίσιο του Horizon και στα πλαίσια της χρηματοδότησης της έρευνας. Υπάρχει ένας κίνδυνος να να θεωρηθεί ότι η αρχή της καινοτομίας έχει ως στόχο κυρίως να μειώσει τη, γραφειοκρατία και να, τη γραφειοκρατία και να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και όχι να λειτουργήσει ως θετικό για τη δημοκρατία. Έχετε ένα, ένα σεμινάριο σχετικά το Δεκέμβριο, αλλά η έμφαση που δίνεται στην, ε, στις επιχειρήσεις μπορεί να δημιουργήσουν μία αντίδραση από πλευράς π.χ. επιχειρήσεων, ε, ε, συνδικάτων, πολιτών. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό. Ευχαριστώ για την Ευρώπη, τη Δημοκρατία και ταυτότητα, ο κ. Μπόκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα στους εκπροσώπους της Φιλανδικής Προεδρίας. Από πλευράς της ομάδας μου θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο επόμενο εξάμεινο για να μπορέσετε να καταλάβετε όλες τις ευαισθησίες που εκφράζει η Επιτροπή μας. Έχω κάποιες ερωτήσεις προς την Υπουργό κυρία Κούλμουνη. Η Προεδρία δήλωσε ότι θέλει εύλογα να επιδιώξει φιλόδοξους στόχους τον μηδενισμό των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακου. Τι, ποιοι μηχανισμοί θα ακολουθηθούν, τι θα κάνετε για να μην έχουμε επιπτώσει στην οικονομία. Επιδοτήσεις. Εμείς βλέπουμε ότι εσείς εμπιστεύεστε την αγορά οι ανανεώσιμες ενέργειες αυτή τη στιγμή αποτελούν τον έναν από τους κλάδους με τη μεγαλύτερη επιδότηση. Μήπως θα έπρεπε και άλλες μορφές ενέργειας να έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Έχω μία ερώτηση και για το Nord Stream 2. Η δήλωση του πρόεδρου της Επιτροπής στον τύπο, όπω όπως αναφέρθηκε στον τύπο, είναι σαφές. Ωστόσο, κατά την άποψή του είναι ένα έργο που θα αυξήσει την ενεργειακή εξάρτηση της Ένωσης. Ποια είναι η άποψή σας σχετικά? Έρευνα. Υπάρχουν προτάσεις από πλευράς Προεδρίας για να μειωθεί η απόκληση μεταξύ των προτάσεων Επιτροπής του Horizon Europe και των θέσεων της Επιτροπής Ήτρε. Μιλήσετε εισαγωγικά, θα ήθελα κάποιε περαιτέρω διευκρινήσει. Μια άλλη ερώτηση, προσανατο... γενικός προσανατολισμός, ε, προβλέπετε κάτι για τον Χάλιβα υπό το φως των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης που εκφράστηκαν. Και μια τελευταία παρήτηση για την Υπουργό κυρία Μαρίν, για το 5G. Όπως ξέρετε, ο Επίτροπος Ασφάλειας δήλωσε ότι ο στόχος είναι μέχρι τέλος του έτους να υπάρχουν κοινά μέσα για την αντιμετώπιση των απειλών ασφάλειας του, των δικτύων 5G. Εδώ είναι σαφές, ε, σαφής η θέση των ε, διαφόρων χωρών. Με, δε, με δεδομένο ότι η Φιλανδία έχει μεγάλη έμφαση στην τεχνολογία αυτή, ποια είναι η άποψη της Προεδρίας σχετικά. Σας ευχαριστώ για την απάντηση που θα δώσετε και σας εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτό το μεγάλο και δύσκολο εξάμεινο της Προεδρίας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις δύο κυρίες που παρουσίασαν το πρόγραμμα της Φιλανδικής Προεδρίας. Δύο ερωτήσεις έχω, αν μου επιτρέπετε. Και θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο προλαλής σας. Γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει εργασίες πάνω σε νέα νομοθετική δέσμη ε, για την αγορά αερίου. Η ερώτησή μου είναι, η Φιλανδική Προεδρία θα οργανώσει κάποιο είδους συζήτηση με τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο θέμα αυτό πριν την οριστικοποίηση της νέας νομοθεσίας. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο αυτό για όλους τους ενδιαφερομένους. Ο συνάδελφος αναφέρθηκε στον αγωγό Nord Stream. Κατά την προηγούμενη θητεία ασχοληθήκαμε με την αναθεώρηση της οδηγίας για το φυσικό αέριο. Αναρωτιέμαι εάν θα επανέλθετε στην διαπραγμάτευση της εντολής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, επαναδιαπραγμάτευση του αγωγού με την Ρωσία. Επίσης, άκουσα ότι γίνονται κάποιες εργασίες για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η ερώτησή μου είναι, σκοπεύετε να κάνετε κάτι στον τομέα αυτόν και θα υπάρξει συντονισμός ε, σε σχέση με τις εργασίες για την ε, οδηγία για τα δικαιώματα του δημιουργού, την οδηγία copyright, διότι αυτό ήταν ιδιαίτερα επίμαχο θέμα κατά την προηγούμενη θητεία, όπως ήταν και τα οπτικοακουστικά μέσα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Από την ΚΟΕ. Καλημέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ο κύριο Μποτέγκα. Και να καλωσορίσω φυσικά και τις υπουργούς θα προεδρεύσετε στο Συμβούλιο, το οποίο φυσικά σημαίνει ότι θα έχετε ιδιαίτερη επιρροή για τις πολιτικές για το επόμενο διάστημα, ε, ε, διάστημα κλειδί για τα ε, κλιματικά και τα κοινωνικά ζητήματα που μας απασχολούν και έχω τρεις συγκεκριμένε ερωτήσεις για το θέμα αυτό, αλλά θα ήθελα καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας κάτι το οποίο βρέθηκε και στο βελγικό τύπο εχθές, ήταν πρώτο θέμα και μάλιστα ήταν και σε μια επιστολή 100 βουλευτών το τον Απρίλιο και είναι κάτι που με απασχολεί ιδιαίτερα. Η επιλογή που έχετε να έχετε ως χορηγό την BMW και μάλιστα σε μια εποχή που για αυτή την κλιματική φιλοδοξία επιλέγετε να συνεργαστείτε με μια αυτοκινητοβιομηχανία η οποία κατηγορείται ότι ε, μπλοκάρισε ή δεν επέτρεψε την ανάπτυξη ε, τεχνολογιών για να περιορίσει τις επιζήμιες ε, συνέπειες κάποιων αερίων καυσίμων θα ήθελα να σας πω ότι για τον κόσμο εδώ έξω αυτά τα πράγματα είναι αδικαιολόγητα. Εσείς ίσως βρείτε, βρείτε κάποια αιτιολόγηση. Τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις λοιπόν για να είμαστε βέβαιοι ότι οι φιλοδοξίες που αναφέρετε εσείς για το κλίμα δεν θα μείνουν κενό γράμμα. Πρώτον, προφανώς ε, συμφωνούμε απολύτως με το στόχο μιας ε, ουδέτερης κλιματικά Ευρώπης ε, μέχρι το 2050 το θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν και τα κατάλληλα μέσα. Θα πρέπει να δοθούν συγκεκριμένα μέσα και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν, ε, χωρίς ε, συγγνώμη, δεσμευτικούς κανόνες προς τις πολυεθνικές, οι οποίες είναι υπεύθυνε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μεγάλο τμήμα της ρήπανσης και των εκπομπών, δεν θα τα καταφέρουμε. Τι είναι αυτό λοιπόν το οποίο δεν θα επέτρεπε σήμερα να προτείνετε τέτοιους κανόνες, να τους προωθήσετε και να τους υπερασπιστείτε και μάλιστα με σθένος. Δεύτερον, Γνωρίζετε ότι καμία οικολογική μετάβαση ε, δεν ε, ε, είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν δεν είναι και κοινωνική μετάβαση. Άκουσα πολλές φορές να αναφέρεστε στην ανταγωνιστικότητα, στην εμπιστοσύνη που δίνεται στις αγορές, αλλά ελάχιστα σχεδόν τίποτα για τους εργαζομένους, για ε, πολύ ισχυρά κοινωνικά μέτρα, τα οποία είναι αυτά που χρειαζόμαστε εάν αυτή η οικολογική μετάβαση ε, δεν θέλουμε να γίνει εις βάρος των εργαζομένων. Και τέλος, το έγγραφο το οποίο μας υποβάλλατε ε, την προηγούμενη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο δίνεται τεράστια σημασία ως προτεραιότητα στα στρατιωτικά ζητήματα και στον πόλεμο. Ξέρετε ότι κάθε ευρώ που δίνεται για στρατιωτικά ζητήματα είναι ένα ευρώ λιγότερο για το κλίμα και τα κοινωνικά ζητήματα. Πώς θεωρείτε ότι είναι συμβατά αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Εάν κάποιος επιθυμεί να πάρει το λόγο, μπορεί να τον πάρει κατά τη διάρκεια του δευτέρου γύρου. Παρακαλώ λοιπόν να πείτε στη γραμματεία αν θέλετε να πάρετε το λόγο, να κάνετε ένα νεύμα. Να στραφώ τώρα στις Υπουργούς για να ακούσουμε τις παρατηρήσεις τους πάνω σε αυτά που άκουσαν μέχρι στιγμής. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις εξαιρετικές ερωτήσεις και παρατηρήσεις σας. Εξαιρετικές παρεμβάσεις. Ε, προσπαθώ να αλλάξω τη σειρά στις απαντήσεις μου. Αρκετοί συντονιστές αναφέρθηκαν στη βιομηχανία. Η κυρία Βίρκουνεν, η κυρία Τόγια αναφέρθηκαν στο θέμα αυτό και η κυρία Δραπάγιοβα αναφέρθηκε στις επενδύσεις, θέμα που σχετίζεται με τη βιομηχανία. Επίσης αναφέρθηκε η αρχή της καινοτομίας, αναφέρθηκε επίσης η βιομηχανία χάλιβα, ε, καθώς και η κοινωνική πτυχή, τα δικαιώματα των εργαζομένων. Σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας αυτές. Να ξεκινήσω λοιπόν από τη βιομηχανία. Είναι απαραίτητο για να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη να έχουμε ε, μια πολυτομιακή οικονομία η οποία να μπορεί να ανταγωνίζεται, να έχουμε ισχυρές εξαγωγές ε, και να μπορέσουμε να ανταγωνιζόμαστε και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό το ανέφερα και στις αρχικές μου παρατηρήσεις. Έχει αλλάξει όμως η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα. Βλέπουν ε, διαφορετικά τα θέματα βιομηχανικής πολιτικής για εμάς τους Ευρωπαίους είναι σημαντικό η βιομηχανία μας να μπορεί να χρησιμοποιεί τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση να γίνεται με τρόπο όσο γίνεται πιο αποτελεσματικό και ευφυή. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και την κυκλική οικονομία. Πιθανότατα να μην χρειαζόμαστε καν λέξη για τα απορρίμματα εάν μπορούμε να επαναχρησιμοποιούμε τα υλικά θα πρέπει να εξετάσουμε και τις κλιματικές μας δράσεις, ε, να γίνουμε οικονομία ουδέτερη ως προς τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε καινοτόμε λύσεις ε, στις ε, δημόσιες αποφάσεις που λαμβάνονται. Πρέπει όμως να συμμετέχουν και οι επιχειρήσεις στη διαδικασία αυτή. Και φυσικά όλα αυτά συνδέονται με το θέμα των δεξιοτήτων. Είναι σημαντικό η εσωτερική αγορά να λειτουργεί καλά, να είμαστε ανταγωνιστικοί και υπάρχουν πολλοί νέοι τομείς που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει βέβαια να λάβουμε υπόψη μας και το θέμα του ιδιωτικού βίου, της προστασίας του ιδιωτικού βίου. Έχουν ληφθεί αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τους πιο σημαντικούς τομείς και γνωρίζουμε βέβαια ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσει είναι η σπονδυλική στήλη της οικονομία μας. Είναι σημαντικές και για την ευημερία των πολιτών. Γι' αυτό είναι σημαντικό η ανάπτυξη της βιομηχανίας ε, να συνοδεύεται από έρευνες. Ακούστηκαν και ερωτήσεις ε, σχετικά με τη βιομηχανική πολιτική συγκεκριμένα τι συγκεκριμένες δράσεις θα αναλάβει το Συμβούλιο. Για παράδειγμα, το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερη ρύθμιση της ε, εσωτερικής αγοράς. Αυτό είναι θέμα πολύ σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας. Να αναφερθώ επίσης στη βιομηχανική στρατηγική μας. Στο πρόγραμμα της Προεδρίας μας αναφέραμε ότι έχουμε μια ολιστική, μια συνολική προσέγγιση, σφαιρική προσέγγιση. Ε, δεν είναι θέμα μόνο βιομηχανικής πολιτικής, είναι ένα οριζόντιο θέμα που αφορά τις εργασίες πολλών ομάδων εργασίας του Συμβουλίου. Ακούστηκαν αρκετές ερωτήσεις για το κλίμα. Πώς θα πετύχουμε τους στόχους που αναφέρουμε στο πρόγραμμά μας. Έχουμε για παράδειγμα τον στόχο για το 2005. Το φθινόπωρο θα συζητήσουμε τα εθνικά ε, ε, ενεργειακά και κλιματικά σχέδια, τα οποία θα είναι τα συγκεκριμένα μέσα ε, που θα χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη. Έτσι πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο, να χαρτογραφήσουμε την κατάσταση στον τομέα αυτών θα λάβουμε στοιχεία και θα πρέπει να προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας ανάλογα με τα στοιχεία που λαμβάνουμε. Τον Σεπτέμβριο θα συζητήσουμε και τα εθνικά σχέδια στο Συμβούλιο. Ακούστηκε επίσης ερώτηση σχετικά με το πώς βλέπουμε την ε, δέσμη μέτρων για το φυσικό αέριο ή ε, πώς βλέπουμε τον αγωγό Nord Stream. Σημαντικό θα είναι όταν πια θα έχει υποβληθεί η δέσμη μέτρων ε, για το φυσικό αέριο να εξετάσουμε και το θέμα του βιοαερίου. Σε αυτήν την ε, δέσμη μέτρων ε, θα επικεντρωθεί μια συζήτηση προσανατολισμού το Δεκέμβριο. Λίγα λόγια επίσης για τον αγωγό Nord Stream και την εντολή. Προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι έχει καταρτισει νομοθεσία για το φυσικό αέριο και κατά τη διάρκεια της Φιλανδικής Προεδρίας ε, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να εφαρμοστεί. Εάν ε, τεθεί στο θεματολόγιο του Συμβουλίου ε, ο αγωγός Nord Stream, η Φιλανδική Προεδρία δεν θα εμποδίσει τη συζήτηση. Επίσης, όσον αφορά τις ε, χαμηλέ εκπομπέ άνθρακα, την, αποδοχή, την κοινωνική αποδοχή του θέματος, ε, τις ερωτήσεις του κυρίου Ποτενκά, φυσικά είναι σημαντικό η ψηφιακή επανάσταση να πραγματοποιηθεί με τρόπο κοινωνικά δίκαιο. Όλο μας ε, το πρόγραμμα βασίζεται σε αυτό. Θέλουμε μια μετάβαση βιώσιμη και κοινωνικά και ε, περιβαλλοντικά. Η ε, Υπουργό Εργασία, η συνάδελφό μου, ίσω να προχωρήσει περισσότερο ει βάθο στα θέματα αυτά. Μας ενδιαφέρει όμως φυσικά ε, να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των πολιτών. Κλείνοντα, ε, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για το πολιετέ ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Η κυρία Βίρκουνεν αναφέρθηκε σε αυτό. Είναι σημαντικό για τη Φιλανδία ε, οι συζητήσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Αυτή είναι μια από τις πιο σημαντικές προτεραιότητές μας. Το ορίζον Ευρώπη είναι σημαντικό θέμα Ήδη είχαμε τριμερείς διαλόγους και θα δούμε πώς θα προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις στη συνέχεια. Σημαντικό είναι πάντως να κλείσει το θέμα αυτό. Και κατόπιν θα προχωρήσουμε σε άλλα ζητήματα στα οποία δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία ακόμη. Κάποιος ρώτησε σχετικά με την αρχή της καινοτομίας. Ο κύριος Νίμιστα αναφέρθηκε στο θέμα αυτό και βέβαια είναι σημαντικό η προσέγγιση αυτή να εφαρμοστεί ήδη κατά την προκατακτική ε, φάση κατάρτισης της νομοθεσίας. Η αρχή της καινοτομίας δεν έρχεται σε αντίθεση με την ε, αρχή της προφύλαξης. Η κλιματική δράση, οι σε, για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, το πρόγραμμα ορίζων, ο στόχος του 25% είναι όλα σημαντικά θέματα και μπορώ να απαντήσω και στην ερώτηση που έχει να κάνει με την ΒΜΒ. Η Προεδρία έχει κάποιες δαπάνες μεταφορών. Όλες οι προεδρίες νομίζω ότι συνάπτουν κάποια συμφωνία με ε, μεγάλες επιχειρήσεις. Η Σουηδική Προεδρία είχε με τη Βόλβο. Η BMW ήταν η μόνη εταιρεία που πληρούσε τις προϋποθέσεις που είχαμε θέσει και γι' αυτό την επιλέξαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κυρία Μαρίν. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω όλους τους ευρωβουλευτές για τις ερωτήσεις. Ε, είναι τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ και να συζητώ αυτά τα τόσο σημαντικά θέματα. Θα αποπειραθώ να απαντήσω ε, σε ό,τι ε, αφορά τις αρμοδιότητές μου. Η κυρία Βιρκουνέν ρώτησε για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σε επίπεδο Συμβουλίου έχουμε ήδη συμφωνήσει σε θέματα που αφορούν ε, το μηχανισμό και πρέπει να βοηθήσουμε να υπάρχουν ε, δράσεις για την ανταγωνιστικότητα. Εδώ η ψηφιοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντική, μας ενδιαφέρει η οικονομία των δεδομένων και όλες οι δράσεις οι οποίες ε, ευνοούν την ψηφιοποίηση. Ε, επίσης, αναφέρθηκε η κλιματική αλλαγή και πώς θα επιτευχθούν οι στέοχοι και εδώ θεωρώ ότι η ψηφιακή ε, τεχνολογία θα μας βοηθήσει. Η κυρία Τόγια ε, αναφέρθηκε στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Εμείς ε, προωθούμε τη σχετική νομοθεσία και το Κέντρο καινοτομία για τα ε, θέματα του κυβερνοχώρου θα αποτελέσει πολύ σημαντική βοήθεια προς τα κράτη-μέλη. Προσπαθούμε να προχωρήσουμε τις διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να συζητήσουμε τον κανονισμό με το Συμβούλιο. Η κυρία Δλαμπάγιοβα ρώτησε για το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη. Θεωρώ ότι το πρόγραμμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, περιλαμβάνει πάρα πολλές δράσεις οι οποίες προωθούν τις ευρωπαϊκές δεξιότητες και πολύ σημαντικούς τομείς. Οι διαπραγματεύσεις ε, με το Κοινοβούλιο ε, θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε για το περιεχόμενο του ε, κανονισμού. Υπάρχουν θέματα βέβαια τα οποία δεν είναι στο δικό μου το χαρτοφυλάκιο, αλλά όταν ε, συμφωνήσουμε για το πρόγραμμα θα προχωρήσουμε ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό. Ο κύριος Νίνιστο, όπως και πολλοί άλλοι, αναφέρθηκαν σε πολύ σημαντικά περιβαλλοντικά και κλιματικά ζητήματα. Είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει μια κοινή αντίληψη με τα κράτη-μέλη για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αυξήσουμε το επίπεδο φιλοδοξίας ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους τη Συμφωνία των Παρισίων. Ε, βεβαίως εδώ χρειάζεται και ε, συνεργασία με το Κοινοβούλιο για να προχωρήσουν τα θέματα, αλλά το επίπεδο φιλοδοξία θα πρέπει να αυξηθεί. Ε, πρόκειται για κάτι ε, το οποίο ε, βρίσκει σύμφωνα πολλά κράτη-μέλη. Ο κύριος Κροσνοντεύσκη αναφέθηκε στο συντονισμό των ψηφιακών θεμάτων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα ψηφιακά ζητήματα θα πρέπει να θεωρούνται σύνολο και όλοι θα πρέπει να βοηθήσουν. Όσον αφορά τα θέματα των πνευματικών δικαιωμάτων και την οδηγία, αυτό είναι κάτι που είναι αρμοδιότητα τη επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμεί, στη διάρκεια τη Προεδρία μα, θέλουμε να συνεχίσουμε τι συζητήσει για τι νέε προκλήσει. Μετά, ο κύριο Μπόρχια ρώτησε για το 5G και την ασφάλειά του. Είναι ξεκάθαρο ότι το 5G είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, ψηφιακές υπηρεσίες, ε, τεχνική, τεχνητή νοημοσύνη και αυτοματοποιημένη οδήγηση είναι θέματα τα οποία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το 5G και πιστεύετε ότι θα πρέπει να διανύμετε στους παρόχους μέχρι το 2020 ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια και οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν να εξελίσσονται βάσει του 5G. Θα πρέπει βέβαια να είναι ασφαλές και να υπάρχει προστασία και ε, συζητώνται στο Συμβούλιο τα θέματα ασφαλείας και προστασίας του 5G. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τις κατευθυντήρες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι πάρα πολύ σημαντικό να κωδικοποιηθούν αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο κράτη-μέλη να καταρτήσουν ένα κατάλογο για τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μπορέσουμε, για παράδειγμα, να ε, παρέχουμε επιστοπίσεις. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν πρέπει να συμμετέχουν ε, στη διαμόρφωση των κανόνων του 5G και στην ανάπτυξή του στη συνέχεια. Ο κύριος Μποτέγκα ρώτησε για τα θέματα του κλίματος, ε, ρώτησε την εφαρμογή των κλιματικών δράσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν φιλόδοξοι στόχοι και να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τους στόχους αυτούς. Ιδάλλως η κλιματική πολιτική δεν θα είναι αποτελεσματική. Ε, αντιλαμβάνομαι την ανησυχία σας και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε και με τα κράτη-μέλη περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και για το ενδιαφέρον που έχετε δείξει. Θα πρέπει να περιορίσω τις παρεμβάσεις όλων για να μπορέσουν να απαντήσουν όλοι για να έχουν χρόνο να απαντήσουν και οι υπουργοί. Ένα λεπτό αν γίνεται. Καρβάλιο. Ευχαριστώ. Κυρίες Υπουργοί, ευχαριστούμε που είστε εδώ. Δύο ερωτήσεις. Κούλμουνη. πίδελτα τα και έρευνα. Μιλήσατε για το ΠΔΠ. Μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση θέλω να θέσω όμως. Η Φιλανδική Προεδρία θα υποστηρίξει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Horizon 2020. Έχουμε 120 δις πρόταση για το Horizon. Και θέλαμε να μας πείτε την άποψή σας για το, την πρότασή μας για το Horizon πάλι. Τι, προγράμματα, τι πρόγραμμα έχει η Προεδρία για την υποστήριξη των δύο πιο σημαντικών καινοτομιών του Horizon Europe. Αποστολές και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας που εξελίσσονται και θέλουν εξ αρχής υποστήριξη. Δεύτερη ερώτηση για την κυρία Πάιν. 5G πολύ σημαντικό για την τεχνολογία. Τι, προγράμματα, τι πρόγραμμα έχει η Προεδρία για να μην μείνει πίσω η Ευρώπη. Μιλήσατε για την ανάγκη ε, να χτίσουμε εμπιστοσύνη με τους ανθρώπους που δεν έχουν να κάνουν ε, με το 5G. Παρακαλώ να τηρείτε το ένα λεπτό Thank you, Madam President, and welcome to both. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε, Κύριε Υπουργοί. Οι κυβερνοεπιθέσει μπορεί να είναι καταστροφικέ. Είδαμε τέτοιες περιπτώσεις πρόσφατα με τεράστιες απώλειες και πιθανές απώλειες. Γι' αυτό καλωσορίζω την σημασία που δίνει η Προεδρία στην κυβερνοασφάλεια. Βλέπω και πόσο σημαντική είναι η τεχνητή νοημοσύνη στο πρόγραμμά σας. Η Φιλανδία ήταν πάντα πρωτοπόρος στα ψηφιακά. Ήσασταν οι πρώτοι που ασχοληθήκατε και με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης συγκεκριμένα. Τι θα κάνετε για να βοηθήσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμορφώσει τεχνολογίες που θα αυξήσουν τα πρότυπα κυβερνό ε, ασφάλειας των επιχειρήσεων. Στην κυρία Κούλμουνη, πώς θα χρησιμοποιήσετε την βελτίωση της τεχνικής νοημοσύνης για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρότι που δυσκολεύονται, παρότι είναι δυναμικές. Πίκανινεν. Ένα λεπτό. Πρόεδρε. Με χαρά σας βλέπω εδώ, κυρίες Υπουργοί. Δύο ερωτήσεις, σύντομες. Η Ευρώπη είχε πει πριν χρόνια ότι θα είμαστε το νούμερο ένα στην παγκόσμια οικονομία. Αποτύχαμε δεν επενδύσαμε επαρκώς. Η ερώτηση είναι η Φιλανδία στην Προεδρία της θα προωθήσει τη συνεργασία για την έρευνα και ανάπτυξη με επιχειρήσεις και άλλους φορείς. Ο στόχος είναι να γίνουν τα νέα ευρήματα το συντομότερο δυνατό προϊόντα που θα πουλούνται, που θα προωθούνται στην αγορά. Μια δεύτερη ερώτηση. Ενέργεια. Τέθηκαν πολλά ερωτήματα για την ενέργεια. Πώς... Τι, τι άποψη έχει την πυρηνική ενέργεια η Φιλανδία. Θα προωθήσετε την ε, εφαρμογή νέων θέσεων εναπόθεση στην Φιλανδία και αλλού. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ερώτηση η δική μου ακολουθεί την ε, ίδια κατεύθυνση. Έχουμε συμφωνήσει μείωση 40% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 30, ε, διότι ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, πέτυχε καλύτερο αποτέλεσμα με τις διαπραγματεύσεις. Η κυρία Φοντερ Λάιεν θέλει 55%. Πώς θα το πετύχουμε αυτό. Η Γερμανία έχει καταλήψει την πυρηνική ενέργεια. Η Γαλλία σκέφτεται μια παράταση της λειτουργίας των πυρηνικών εργαστηρίων. Η Φιλανδία έχει ήδη τέσσερις και χτίζει άλλη μία εγκατάσταση με ρωσική υποστήριξη. Βλέπετε εσείς κάποια εναλλακτική λύση για να πετύχουμε τους στόχους μας όσον αφορά το κλίμα. Ποια είναι η θέση της Φιλανδίας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πραγματικά ήσασταν υπόδειγμα όσον αφορά το χρόνο ομιλίας. Ο κύριος Μπλος, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, ε, κυρίες Υπουργοί. Καταρχάς, ε, συγχαρητήρια που θέσατε την ε, θέρμανση του πλανήτη ε, και το κλίμα στον πυρήνα των εργασιών της προεδρία σας καθώς και το φιλόδοξο στόχο του να έχετε μια ε, κλιματικά ουδέτερη Φιλανδία μέχρι το 2035. Ανήκω σε μια γενιά νέων ανθρώπων που φοβούμαστε ότι η κλιματική κρίση θα καθορίσει τη ζωή μας και πρέπει να αναλάβουμε δράσεις ε, τώρα αμέσως. Από τη Βάδη Βιρτεμβέργη προέρχομαι ε, και το Συμβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ε, πολιτική ώστε να γίνουμε ουδέτεροι ως προς το κλίμα μέχρι το 2050 και να μειώσουμε τις ε, εκπομπές ε, κατά 50% μέχρι το 2030. Δύο ερωτήσεις λοιπόν. Εσείς τι θεωρείτε ότι είναι πιο σημαντικό για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς στη βιομηχανική πολιτική. Δεύτερον, η Κομισιόν και το Συμβούλιο πώς πρέπει να αλλάξουν ε, τους ισχύοντε τομεακού στόχου ε, και τρίτον, ε, ποιε πιστεύετε ότι είναι οι εύκολε λύσει, οι άμεσε λύσει όσον αφορά την κλιματική κρίση, τι μπορούμε να πετύχουμε γρήγορα, διότι πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Να δω πού βρισκόμαστε, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Γκάιερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Χάλιβα. Ε, πρέπει να ε, αγωνιστεί σε καιρούς ε, πλεονασμάτων ε, σε όλο τον κόσμο και τα μέτρα προστασίας που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν φανεί ανεπαρκή μέχρι τώρα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η Φιλανδική Προεδρία πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει το θέμα. Ε, σκέφτεστε να έχετε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τους τομείς κλειδιά για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπουχάιτ, παρακαλώ. Καλημέρα και από μένα. Σύμφωνα με ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, Παραγωγών ε, Μηχανών φαίνεται ότι ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας ε, οι τιμές ρεύματος είναι υπερβολικά υψηλές ε, ενώ από την άλλη έχουμε την ε, αυτοκινητοβιομηχανία ως κινητήρα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Πώς μπορούμε να έχουμε μείωση των εκπομπών χωρίς να έχουμε μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων και πώς μπορούμε να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για τις βιομηχανίες μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σκίτεταν, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ερώτησή μας απευθύνεται στην κυρία Μαρίν. Ε, ήθελα πιο συγκεκριμένα στοιχεία όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια. Βλέπουμε ότι βρυδικέ ε, δράσει ε, όπω είναι οι κυβερνοεπιθέσει ε, και η παρέμβαση σε εκλογέ επηρεάζουν τη διαμόρφωση πολιτική, αποδυναμώνουν την κοινωνία και υπονομεύουν την ενότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά το γεγονό ότι είναι ε, επίγον το θέμα, ε, τα δύο θεσμικά μα όργανα δεν έχουν πετύχει ε, συμφωνία όσον αφορά ευρωπαϊκό σχέδιο για την κυβερνοασφάλεια και το βασικό πρόβλημα είναι η λειτουργία του κέντρου, η χρηματοδότηση και το νομικό καθεστώς. Είπατε ότι είσαστε τεθμένοι να συνεχίσετε τις διαπραγματεύσει και αρκετοί συνάδελφοι ανέφεραν πόσο επίγον είναι το θέμα. Η ερώτησή μου είναι η εξή τι πιθανότητες έχει το Συμβούλιο να λάβει νέα εντολή διαπραγμάτευσης με βάση τη Συμβουλή της Νομικής Υπηρεσίας του Συμβουλίου πάνω στο επίγον αυτό θέμα. Και τι πιθανότητες υπάρχουν για συμφωνία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέχρι το τέλος ε, της ε, Φιλανδικής Προεδρίας. Με άλλα λόγια, θα ήθελα το χρονοδιάγραμμα για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Στέγκρουτ. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριες Υπουργοί, τα, οι κλιματικοί στόχοι όσον αφορά ε, το, τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ήταν πολύ αργές και δέκα χρόνια έχουμε στη διάθεσή μας, σε 25 χρόνια εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα και γνωρίζω πολύ καλά ποιες είναι οι προϋποθέσεις ε, στην αγορά. Γνωρίζω επίσης ότι είναι ε, πολύ χρονοβόρες και ακριβές ε, οι σχετικές επενδύσεις. Δέκα χρόνια στο πλαίσιο αυτό δεν είναι τίποτα. Γνωρίζω και πολλά για τον ανταγωνισμό. Γνωρίζω ότι για μεγάλο μέρος ε, της βιομηχανίας η ανταγωνιστικότητα βασίζεται στις χαμηλές τιμές. όλα αυτά θα δυσκολέψουν ακόμη την κατάσταση. Ε, ως οικονομολόγος ε, βλέπω να βρισκόμαστε σε ε, κυκλική φάση χαμηλής ανάπτυξης. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ χωρί μικρόφωνο. Πρέπει να μιλήσετε στο μικρόφωνο, γιατί αλλιώ ε, δεν μπορώ να καταλάβω τι λέτε. Δεν σα ακούω. Sorry, eh, Η ερώτησή μου λοιπόν είναι οι φιλόδοξοι κλιματικοί στόχοι θα μπορέσουν να διατηρηθούν σε περίοδο ε, χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης ή θα κάνουμε εκπτώσεις στις φιλοδοξίες μας. Ευχαριστώ. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Καλβέθ νιώθει τώρα. Καταρχάς, ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε δύο γυναίκες ε, ε, σε τομείς που συνήθως κυριαρχούν οι άντρες και να ευχηθώ ότι καλύτερο για τη Φιλανδική Προεδρία. Δύο ερωτήσεις, μία για το ορίζον και μία για το ψηφιακό θεματολόγιο. Όσον αφορά το ορίζον, αν ε, κατάλαβα καλά, συμφωνείτε και συμφωνούμε και εμείς ότι πρέπει να διαθέσουμε περισσότερους πόρους για την έρευνα και την καινοτομία, αλλά θα πρέπει να γίνει αυτό και με περισσότερη διεθνή συνεργασία και συνέργειες. Ε, να επιμένω στην ερώτηση, ε, εσείς υποστηρίζετε την αύξηση των 120 δισεκατομμυρίων ευρώ που έγιναν από την Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ορίζον και επίσης για το παράδειγμα 4 για διατομιακή και συνεργασία και συνεργασία μεταξύ χωρών για το ορίζον ε, Ευρώπη. Και επίσης για το ψηφιακό ε, θεματολόγιο, ποια είναι η, η άποψή σας για την κοινή φορολόγηση ε, για τις ε, πολυεθνικές επιχειρήσεις και επίσης για τεχνολογικές ε, πλατφόρμες και τις συνθήκες εργασίας. Και επειδή μου άρεσε, είπατε ότι χρεια... θέλουμε μια πολιτική η οποία θα έχει στο επίκεντρο τους ανθρώπους. Θα υπάρξει και διάκριση λόγω φίλων, φίλου στην τεχνητή νοημοσύνη. Ευχαριστώ. Η κυρία Σόλης Περέδ. No, you didn't uh, raise your... No, it's okay then. Δεν θέλετε το λόγο. Εντάξει, δεν πειράζει. Η κυρία Βάιθ. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Η ερώτησή μου κυρίως απευθύνεται προς εσάς, ε, κυρία Κούλμονη. Uh, Το πρόγραμμα της Προεδρίας ε, που ε, μας παρουσιάσατε θέλει να ενισχύσει την κινητικότητα των εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει και να διευκολύνει και την έλευση ε, εξειδικευμένου προσωπικού από τρίτες χώρες. Στη Δανία έχουμε 7.000 ανεπιτυχείς προσλήψεις κάθε χρόνο και αυτό είναι πρόβλημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας στην Ευρωπαϊκή η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξή. Τι δράσεις ε, ε, πιστεύετε ότι θα πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ε, διευκολύνει την ε, κινητικότητα των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρόπε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να θέσω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις για την πυρηνική ενέργεια. Όπως γνωρίζετε η χώρα μου κλείνει ε, πυρηνικά εργοστάσια. Το 2012 έγινε ένα δημοψήφισμα το οποίο ε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να σταματήσει η χρήση πυρηνικής ενέργειας. Αλλά δίπλα στα σύνορα η Λευκορωσία ε, ολοκληρώνει το πυρηνικό της εργοστάσιο στο Όστροβιες. Ε, έχουν καταλήξει και σκοπεύουν ε, να ξεκινήσουν τις εργασίες έγινε και ε, μια δοκιμασία αντοχής ε, και βάσει των αποτελεσμάτων φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις ε, στο εργοστάσιο αυτό. Το θέμα είναι τι σκοπεύετε να κάνετε για να μην επιτρέψετε στη Λευκορωσία να προωθήσει νέα πυρηνικά εργοστάσια χωρίς να αντιμετωπίζει και τα προβλήματα και τις ελλείψεις. Αυτό είναι πρόβλημα όχι μόνο για τη Λιθουανία αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Γεωργίου παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τις ε, δύο υπουργούς για τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους και εύχομαι κάθε καλό στην Φιλανδική Προεδρία προς την κυρία Κουλμουνή η οποία υπογράμμισε ότι στις προτεραιότητες της Προεδρίας είναι η Ενεργειακή Ένωση και η ενίσχυση της ασφάλειας. Τρία ερωτήματα. Πώς διασφαλίζεται αυτή η ενεργειακή ασφάλεια όταν αυτή τη στιγμή η Τουρκία κατά τρόπον παράνομων διεξαγάγει γεωτρήσεις στην Κυπριακή Ναό και έχουμε ένα συμβούλιο το οποίο δυστυχώ εγκρίνει κυρώσει κατώτερε των περιστάσεων. Και δεύτερον, εάν η Φιλανδική Προεδρία σκοπεύει να αναλάβει νέε πρωτοβουλίε οι οποίε να εξαναγκάζουν την Τουρκία να προσέλθει σε παραγωγικέ συνομιλίε για επίλυση του Κυπριακού στη βάση του πλαισίου Κουτέρε. Τρίτον, μιλήσατε για την ενεργειακή φτώχεια. Αναφέρομαι εγώ στην ενεργειακή φτώχεια, όταν είναι στου τέσσερι πολίτε τη Ένωση δυστυχώ βασανίζονται από αυτό το πράγμα, εάν σκοπεύετε να καταθέσετε κάποιον ολοκληρωμένο σχέδιο για στήριξη αυτή τη ε, προσπάθεια. Και το τελευταίο, επαναλαμβάνω πολύ σύντομα ένα ερώτημα το οποίο θεωρώ ότι δεν απαντήθηκε. Στηρίζεστε από την BMW σε ό,τι αφορά στην Προεδρία σας. Θεωρείτε ότι αυτό είναι διοντολογικά ορθό. Okay. Ωραία. Ο κύριος Έγκλαντ και στη συνέχεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέροντα θέματα θέσατε. Κυβερνοασφάλεια για παράδειγμα που η Βρετανία το θεωρεί ως ε, μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη χώρα. Στον προϋπολογισμό του ΠΙΔΕΛΤΑ ΔΕΛΤΑΠ. αυτό ότι ο προπολογισμό για το ΔΠΠ ΔΕΛΤΑΠ περιλαμβάνει και συνεισφορά της Βρετανίας. Ζωρίνιο. Ευχαριστώ. Να καλωσορίσω και εγώ την Φιλανδική Προεδρία και να απευθύνω μία ερώτηση για την ενεργειακή φιλοδοξία και την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Η νέα πρόεδρος της Επιτροπής πρότεινε έναν νέο ευρωπαϊκό Green Deal. Ταυτόχρονα ωστόσο οι πληροφορίες που παίρνουμε από τα εθνικά προγράμματα των κρατών μελών για την συνέργεια στο κλίμα, όπως τουλάχιστον είπαν οι επίτροποι Κανιέτη και δείχνουν ότι τα εθνικά προγράμματα δεν επιτρέπουν να φτάσουμε στους στόχους που έχουμε θέσει. Πώς, θα, πώς προτίθεται η Προεδρία να παροτρύνει τα κράτη-μέλη ώστε να εφαρμοστεί η έκθεση για τη διακυβέρνηση της ενέργειας και να επιτευχθούν οι στόχοι της ενεργειακής ε, αποτελεσματικότητας και των ανανεώσεων. Ευχαριστώ.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 πρέπει να είναι πρωτοπόρος στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Μιλάμε για μια μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ρήπων. Αυτά όλα όμως πρέπει να γίνονται με σεβασμό του ανθρώπου και με στόχο τη βελτίωση της ε, ζωής του. Εμείς θα έπρεπε, θέλουμε ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Λεγγύης για τη μετάβαση αυτή. Προέρχομαι από μια χώρα, μια περιοχή στην Πολωνία, τη Σιλεσία, που έχει μεγάλη σύνδεση με τον άνθρακα. Θα αναλάβετε αυτή την πρωτοβουλία. Μιλάμε για ε, φτώχεια, έλλειψη ενέργεια, ενέργειας. Δεν μιλάμε επαρκώς για ανθρώπους που έχουν που είναι ενεργειακά φτωχοί. Όταν μιλάμε για την αλλαγή του κλίματος, ε, ξεχνάμε μερικές φορές ότι αυτό σημαίνει αλλαγή του κόστους της ενέργειας για ανθρώπους που είναι φτωχοί. Πώς θα αντιμετωπίσετε και την κερδοσκοπία στις τιμές των, ε, των εκπομπών ρήπων. Ευχαριστώ. Κύριος Αντινόλφη. Πρόεδρε, μία ερώτηση για την ψηφιακή ασφάλεια. Καλό είναι να θυμίσουμε ότι στην Ένωση υπάρχουν 4.000 προσπάθειες ε, ψηφιακής απάτης την ημέρα. Σε κάποια κράτη-μέλη το 50% των αδικημάτων που διαπράττονται έχουν ε, είναι χαρακτήρα, γίνονται μέσω ίντερνετ. Άρα ε, Εξού και η σημασία της κυβερνοασφάλειας. Αυτά που είπατε μέχρι τώρα είναι ενδιαφέροντα για όλους. Δείξατε την ε, σημασία, τη σημασία που δίνετε στην προβληματική αυτή. Όλα αυτά όμως έχουν σημασία αν έχουμε κονδύλια σχετικά και για την ε, κυβερνοασφάλεια και στην, για την ετόπιση της κυβερνοασφάλειας από την Europol. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε, λέει η κυρία Τουσάν. Κυρία Υπουργέ, δείξετε βούληση, αλλά μέχρι τώρα κανένα κράτος μέλος ούτε η Ένωση δεν σέφονται τη συμφωνία του Παρισιού. Η δέσμευση μείωσης κατά 50-55% των εκπομπών ε, στην πράξη είναι ε, πολύ μακριά από τους στόχους. Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ωστόσο είναι γνωστά. Γιατί δεν τα υλοποιείται. Κάθε χρόνο η Ένωση δαπανά 4 δις ευρώ άμεσων ενισχύσεων στις ορυκτές πηγές ενέργειας. Για να μην μιλήσω για πολύ περισσότερα δηλαδή από ό,τι αυτά που δίνεται για την έρευνα και ανάπτυξη. Στην ουσία τα χρήματα αυτά πηγαίνουν στις μεγάλες επιχειρήσεις με σκανδαλώδη τρόπο. Δεν μπορούσαμε τα χρήματα αυτά να τα δώσουμε για την, μετάβαση, για την οικολογική μετάβαση. Αυτή τη στιγμή η ΣΕΛ, η ΤΟΤΑΛ αντιμετωπίζουν ε, αγωγές από Ευρωπαίους πολίτες για τις δράσεις τους κατά, ε, κατά του κλίματος και η Ένωση δεν κάνει τίποτα. Τίποτα δεν υπάρχει επιτάπητος για να αντιμετωπίσουμε την κρίση στο κλίμα. Θα χρησιμοποιήσετε κύριε Υπουργέ το θέμα των επενδύσεων στο δημόσιο και της νομικής ρύθμισης στον ιδιωτικό τομέα για την αντιμετώπιση της κρίσης στον πλανήτη μας. Επόμενος ομιλητής. Γκονζάλες Κασάρες. Ο κύριος Γκονζάλες Κασάρες, συγγνώμη. Θα βελτιωθώ, θα βελτιωθώ. Εντάξει, το δεχόμαστε. Καλώ ήρθατε κύριε Υπουργοί στην Επιτροπή μας και ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ξέρουμε ότι η Φιλανδική Προεδρία έχει σαφή δέσμευση για τον αγώνα για το κλίμα. Στην προηγούμενη θητεία συζητήσαμε πολλά για το κλίμα, πέρασε μία οδηγία για τα ανανεώσιμα. Οι στόχοι αυτοί ωστόσο ε, δεν έχουν να ευθυγραμμιστεί με τη συμφωνία του Παρισιού. Επίσης, πολλές χώρες έχουν επιφυλάξεις, ιδίως ό,τι αφορά την ενεργειακή μετάβαση. Η Προεδρία σας έχει σαφείς στόχους και υποχρεώσεις να αντιμετωπίσει τις αλλαγές αυτές. Πώς θα εξασφαλίσετε από τη θέση σας ότι οι, τα εθνικά προγράμματα, τα οριστικά εθνικά προγράμματα για την ενέργεια και το κλίμα θα καλύψουν τα κενά που έχουν για να επιτύχουν πραγματικά τους στόχους που έχουμε θέσει. Θα εξετάσετε τους επόμενους μήνες το ενδεχόμενο να αυξήσετε τους στόχους στην, ε, στα ανανεώσιμα και την ε, από ενεργειακή ασφάλεια. Επίσης πρέπει μακροπρόθεσμα να δεσμεύσουμε μια ουσιαστική στρατηγική. Και μια ακόμα ερώτηση. Σε τι θα στηριστείτε για να εξασφαλίσετε ότι το επιφυλακτικό Συμβούλιο θα υποστηρίξει την κλιματική ουδετερότητα το 2050. Ευχαριστώ. Ας δούμε. Ο κύριος παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε αναθέσει ε, μελέτη σχετικά με τους κινδύνους ε, για την υγεία του δικτύου 5G που ε, θα πρέπει να γίνει από ανεξάρτητους επιστήμονες. Δεύτερη ερώτηση. Το αποτέλεσμα αυτής της μελέτης θα υπάρξουν πριν την επέκταση του δικτύου. Και ερώτηση για τη βιομηχανία Χάλιβα. Ε, μιλήσατε για τις δυσκολίες ε, της βιομηχανίας αυτής. Εάν θέλουμε να περάσουμε όμως σε μια πράσινη βιομηχανία, αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς ε, την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, τι προσπάθειες θα, καταλάβετε, θα καταβάλλετε στο θέμα αυτό. Ο κύριος Τοπισόφσκι. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Οι προλαλήσαντες μίλησαν για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, μίλησαν για τη βιομηχανία μας. Η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει αναφερθεί στο θέμα της φορολογίας προϊόντων και επιχειρήσεων που θα εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν δεν πληρούν κάποιες περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Είναι ενδιαφέρουσα η ιδέα αυτή. Ξέρω ότι δεν είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί, διότι φορολογούμε υπερβολικά τους εαυτούς μας και κατόπιν εισάγουμε προϊόντα με τεράστιο οικολογικό αποτύπωμα. Έτσι λοιπόν ε, υπονομεύουμε τον εαυτό μας. Αναρωτιέμαι εάν θα υιοθετήσετε την ιδέα αυτή της Πρόεδρου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φούλσανγκ. Ε, Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τις υπουργού που έθεσαν τόσο ψηλά στο θεματολόγιο το θέμα ε, του κλίματος. Η ερώτησή μου συνδέεται με την ερώτηση του, μου, του συναδέλφου μου Κονσάλες Καθάρης ε, σχετικά με το πώς μπορεί να επιτευχθεί η συμφωνία όσον αφορά τις φιλοδοξίες μας αυτές ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τον προηγούμενο μήνα το Συμβούλιο δεν μπορούσε να συμφωνήσει ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ουδέτερη ως προς τις εκπομπές το 2050. Αναρωτιέμαι ε, πώς ε, σκοπεύετε να επανεκκινήσετε αυτές τις συζητήσεις ώστε να συμφωνήσουν όλοι με τη στρατηγική αυτή και πώς προβλέπετε να πετύχετε συμφωνία πώς ε, προβλέπετε να πετύχετε τη συμφωνία όλων των χωρών. Θα αποζημιώσετε κάποιες χώρες που θα πρέπει να κάνουν σημαντικές μετατροπές. Πώς βλέπετε την όλη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κέλλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι κάθε επιτυχία στη Φιλανδική Προεδρία. Νομίζω ότι ε, πολλές φορές έχουμε υπερβολικά πολλές ε, προσδοκίες από ε, κάθε Προεδρία, αλλά είναι φιλόδοξη η στόχη σας. Πιστεύω όμως ότι θα τους πετύχετε. Θα πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τα καύσιμα, τον άνθρακα για παράδειγμα, η Φιλανδική Προεδρία πώς θα φροντίσει να είναι δίκαιη η μετάβαση μετά τη συζήτηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, ώστε να μην μείνουν πίσω κάποιες ομάδες του πληθυσμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κριστόφ τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου καταρχάς να ευχαριστήσω τις Υπουργούς για τις αναλυτικές πληροφορίες που μας έδωσαν. Οι κυβερνοεπιθέσεις και η κλοπή ψηφιακής ταυτότητας είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Στη Βουλγαρία μέχρι σήμερα 5 εκατομμύρια Βούλγαροι πολίτες ε, έχασαν, ε, ε, ε, έπεσαν θύματα κλοπής των ψηφιακών του στοιχείων από την Υπηρεσία Φόρου Εισοδήματος. Το Συμβούλιο ενέκρινε ένα πλαίσιο για, την, για κυρώσεις και μέτρα αντίδρασης για τις κυβερνοεπιθέσεις. Τι άποψη έχετε για την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων. Και μία ακόμα ερώτηση. Αναφέρεστε ε, σε δεντολογικό τρόπο εισαγωγής ε, της ψηφιακής οικονομίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Ε, καλωσορίζω την ιδέα σας μεν, αλλά πώς θα το καταφέρετε αυτό, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο ε, θα συμβεί και μετά από την Προεδρία σας. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάν. Κυρία Χάν. The Then uh, yeah. Η κυρία Dowding. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω ότι η Φιλανδική Προεδρία για το μέλλον των εταιρικών συμπράξεων υγείας και έρευνας και ανάπτυξης, διότι ε, πρέπει να γίνουν αξιολογήσει επιπτώσεων εντός ολίγου. Από άποψη πρασίνων θα πρέπει να υπάρχει κοινωνικός αντίκτυπος και θα πρέπει να συμβάλλουν και στην εφαρμογή των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Υπάρχουν ε, δύο εταιρικέ συμπράξει υγεία ε, και έρευνα και ανάπτυξη. Είναι ένα πρόγραμμα για τις ε, κλινικές δοκιμές ε, μεταξύ ευρωπαϊκών και τρίτων χωρών αναπτυσσόμενων. Αυτό υποτίθεται ότι θα βοηθήσει και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Και η δεύτερη εταιρική σύμπραξη υποτίθεται ότι θα επιτύχει την πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα. Και εκεί υπήρχαν επικρίσεις από πολλές πλευρές. Οι επίσημες αξιολογήσεις επιρογνωμόνων έχουν αμφισβητήσει την δυνατότητα να υπάρχει κάποιος κοινωνικός αντίκτυπος και επομένω υπάρχει ανάγκη για σοβαρή μεταρρύθμιση και ανάγκες ε, δημόσιας υγείας ε, για να υπάρχουν κατάλληλες προτεραιότητες ώστε να φροντίσουμε να υπάρχουν διατάξεις για προσβασιμότητα ε, και προσιτά φάρμακα από αυτές τις συμπράξεις για την έρευνα και ανάπτυξη τι άποψη έχει η Προεδρία για αυτέ τι μελλοντικέ συμπράξει και τι μεταρρυθμίσει και κυρίω για το πώ μπορούμε να εγγυηθούμε κοινωνικό αντίκτυπο και να υπάρχει και συμβολή στου στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη και πώ μπορούμε να το εξασφαλίσουμε αυτό στι μελλοντικέ συμπράξει. Ε, παρακαλώ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Οι υπόλοιποι ομιλητέ είναι από του σοσιαλιστέ και δημοκράτε και θα ήθελα να ρωτήσω από τι υπόλοιπε πολιτικέ ομάδε αν έχουμε παραβλέψει κάποιον ο κύριος Κουμπίλιους, η κυρία Βίρκουνεν. Άλλο ναι. ε, Άλλος κανείς. Ο κύριος Κουμπίλιους, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια στη Φιλανδική Προεδρία. Θα ήθελα να επιστρέψω σε κάποιες ερωτήσεις. Στο πρόγραμμα της Προεδρίας θέτετε πολύ σαφείς δεσμεύσεις και σας παραθέτω. Μια συνολική μακροπρόθεσμη στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα και επίσης ότι ο στόχος μας θα πρέπει να είναι η Ευρώπη να είναι παγκόσμιο ηγέτης της ψηφιακή οικονομίας. Και η ερώτησή μου είναι τι θα κάνετε ακριβώς στη διάρκεια της προεδρία σας. Τι έγγραφα θα προτείνετε αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλες προκλήσεις ανταγωνιστικότητας και προσπαθούμε να γίνουμε πρωτοπόροι στην ψηφιακή οικονομία παγκοσμίω, αλλά τι θα κάνουμε αν βρεθούμε να καθυστερούμε τόσο πολύ ε, σε σχέση με τις μεγάλους ηγέτες, τη Microsoft, την Google, την Amazon, είχαμε και την Nokia στη Φιλανδία, αλλά ε, πλέον πάει. Ε, τι προβλέπετε λοιπόν για το μέλλον για αυτά τα θέματα. Ωραία, ευχαριστώ. Η κυρία Καλιούραντ. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις και να σας ευχηθώ ότι καλύτερο για την Προεδρία σας. Δεν θα επαναλάβω ερωτήσεις που αφορούν την κυβερνοασφάλεια που έθεσαν οι συνάδελφοι. Πολύ ευχαρίστω να ακούσω τι έχετε να πείτε επί του θέματο. Η ερώτησή μου αφορά την ε, ε, ταυτοποίηση στο διαδίκτυο. Εγώ είμαι από την Εστονία και επομένω έχω το προνόμιο να μπορώ να απολαμβάνω ψηφιακέ υπηρεσίε διαδικτυακέ υπηρεσίε εδώ και χρόνια. Και ξέρουμε ότι η βάση για τι ηλεκτρονικέ υπηρεσίε, τι διαδικτυακέ υπηρεσίε και νέα αγορά είναι η δυνατότητα ταυτοποίηση στο διαδίκτυο. Και εδώ φυσικά η Ευρώπη υστερεί. Έχουμε χώρε με διαφορετικά συστήματα καθεμία. Επομένως, η ερώτησή μου είναι τι μπορείτε να κάνετε και τι μπορεί να κάνει η Φιλανδική Προεδρία ώστε να υπάρχει ψηφιακή αναγνώριση ταυτότητας στο διαδίκτυο με υψηλά πρότυπα ασφαλεία και να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης και διάθεση σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Βίρκουνεν. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ξέρω ότι Είμαστε στο δεύτερο γύρο και ξαναπαίρνω το λόγο, αλλά θα ήθελα να επαναλάβω την πρώτη με ερώτηση για το δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί νομίζω ότι δεν λάβαμε απάντηση ε, επ' αυτού. Κυρία Κουλμούνη, μας είπε ότι είναι το πιο σημαντικό θέμα για την ε, Φιλανδική Προεδρία να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για το πολιετές, αλλά φυσικά είναι και πολύ σημαντικό, αλλά και το περιεχόμενο είναι πολύ σημαντικό και το τι περιλαμβάνει αυτή η απόφαση. Και η Υπουργό Μαρίν μας είπε ότι η Φιλανδία πιέζει και είναι θέμα εθνικής πολιτικής και δεν μπορώ να συμφωνήσω. Είστε προεδρεύον τώρα του Συμβουλίου και είναι πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο να ξέρουμε και τι στάση θα τηρήσετε εσείς για τις διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, κυρίως για το Connecting Europe Facility, το Horizon Ευρώπη. Ε, είναι προγράμματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την ανταγωνιστικότητά μας και μας ενδιαφέρουν ε, και τη βιομηχανική κοινότητα. Επομένω, θα ήθελα να ξέρω λίγο περισσότερα για τη θέση τη Φιλανδία για αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ που ε, αναφέρετε και πάλι το θέμα, ο κύριος Χάισελ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Με χαρά άκουσα από την Υπουργό Κουλμίνη ότι επαφείται στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν για το ενεργειακό μείγμα. Τώρα θα μιλήσω στη μητρική μου. Είναι σαφές ότι τα ορυκτά καύσιμα δεν θα μπορέσουν να παραμείνουν στο ενεργειακό μείγμα. Η ερώτησή μου τώρα είναι η πυρηνική ενέργεια. Είναι μια πηγή ενέργειας χωρίς χρήση άνθρακα, αλλά υπάρχει πολύ λίγη ε, διάθεση και προθυμία για χρήση της πυρηνικής ενέργειας, παρά το γεγονός ότι οι επιστημονικές ενδείξεις ε, ποικίλουν, κυρίως όσον αφορά τους κινδύνους ασφαλείας. Ε, η ερώτησή μου είναι πώς βλέπετε εσείς το μέλλον της πυρηνικής ενέργειας κυρίως στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, διότι ε, εκεί χρησιμοποιούσαν ορικά καύσιμα, συγγνώμη, μετά πέρασαν στην πυρηνική ενέργεια. Χωρίς την πυρηνική ενέργεια δεν θα είναι σε θέση να επιτύχουν το στόχο των χαμηλών ε, ε, εκπομπών, πολλό δε μάλλον των μηδενικών. Ευχαριστώ πολύ και τελευταίοι τέσσερις ομιλητές από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, η κυρία Μάρκες. Ναι. Ευχαριστώ. Και εγώ να συγχαρώ τη Φιλανδική Προεδρία για το πρόγραμμά της και τις υπουργού που είναι εδώ σήμερα. Δύο σύντομες ερωτήσεις. Με ικανοποίησε ιδιαίτερα το ότι θέσατε του, την ψηφιακή ατζέντα ως προτεραιότητα όχι μόνο από την οπτική του, της ανταγωνιστικότητας αλλά και της συμπερίληψης. Η ερώτησή μου είναι η εξή. Η φιλανδική κυβέρνηση, από ό,τι ξέρω, όρισε ως στόχο να δώσει σε ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της κατάρτιση στον τομέα της ε, τεχνητής νοημοσύνης απλούς πολίτες, όχι ειδικού. Με βάση την εμπειρία σας μπορούμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο στην Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες στο τομέα αυτό είναι απαραίτητες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και το φόβο των αλλαγών μεταξύ του πληθυσμού. Η δεύτερη ερώτηση, το έλεγε και ο αισθανός συνάδελφος, την διαλειτουργικότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών μηχανογραφικών συστημάτων και της ασφαλούς ταυτοποίησης που παρά τα πολλά πιλωτικά έργα που έχουν ξεκινήσει συνιστούν εμπόδιο για την ύπαρξη μιας ενιαίας, ε, πραγματικά ενιαίας αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών. Τι θα κάνετε σχετικά. Η κυρία Μαλντονάντο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και ευχαριστώ της Υπουργού, συγχαρητήρια και την παιδεία σας. Διαβάσαμε το πρόγραμμα που μας παρουσιάσατε και το κείμενό σας και πρέπει να σας πω ότι σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ με το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως στον ψηφιακό τομέα. Υπάρχει κάπου που αναφέρεστε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα σταθώ σε αυτό. Θέλω να ρωτήσω ποιος είναι ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά την άποψή σας στο πρόγραμμα Intel Europe πάνω από ένα δις πόρων. Πώς, με τι συγκεκριμένες δράσεις υλοποιούνται αυτά. Πώς μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δημιουργήσουν μια ψηφιακή ευρωπαϊκή ατζέντα με μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και καλύτερη δυνατότητα δημιουργίας θέσεων εργασίας. Δεύτερη ερώτηση. Ασφάλεια καταναλωτών. Τι συγκεκριμένα μέτρα πιστεύετε ότι πρέπει να υλοποιηθεί από την Προεδρία σε ό,τι αφορά τον τομέα αυτό. Φριτσόν. Κυρίες Υπουργοί, ευχαριστούμε για τις παρατηρήσεις σας. Εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Στο πρόγραμμά σα υπογραμμίσατε τη σπουδαιότητα της έρευνα και της καινοτομία. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, κλίμα, λαϊκισμός, απαιτεί σε κάθε περίπτωση η Ευρώπη να είναι πρωτοπόρο στην έρευνα και την ανάπτυξη. Είναι σαφές ότι το Horizon Europe θα είναι σημαντικό εργαλείο. Πρέπει να θέσουμε σωστές προτεραιότητες προωθώντας και την ισότητα των φύλων και στην έρευνα. Το πρόγραμμα έρευνας πρέπει να έχει ως ορόσημο τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΙΕ. Μια άλλη ερώτηση. Σημαντικό είναι να εξασφαλίσουν οι χώρες της Ένωσης την ελευθερία, την ακαδημαϊκή ελευθερία. Αν αυτό δεν συμβαίνει σε όλα τα κράτη-μέλη, είναι σαφέ ότι οι χώρε αυτέ δεν θα έπρεπε να μπορούν να μετέχουν στο νέο πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Τέλεια. Χόμπς, τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ που ήρθατε να μας πείτε το πρόγραμμά σας και να απαντήσετε σε ερωτήσεις μας. Για τη βιομηχανία θέλω να ρωτήσω πυλώνας της οικονομίας με ένα στις πέντε θέσεις εργασία και είναι υπεύθυνη για μεγάλο κομμάτι των εξαγωγών και κινητήρια δύναμη για την έρευνα στην Ευρώπη. Έχουμε μπροστά μας την πρόκληση να μετατρέψουμε τη βιομηχανία σε κάτι πιο βιώσιμο και με βάση τη γνώση, καθώς και για παραγωγή με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Αυτό αποτελεί, απαιτεί νέες προκλήσεις. Και αυτό είναι το θέμα του εργασιακού ε, του χάσματος. Εργαζόμενους που έχουν πολλές ε, γνώσεις και η ερώτησή μου είναι ποιες είναι οι προτεραιότητες της Προεδρίας ό,τι αφορά την πορεία που θα πάρει η Ευρωπαϊκή Οργανία και οι συναφείς θέσεις εργασίας εν ώψη του μέλλοντος ιδίω από την οπτική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες διαχείρισης των πόρων αυτών και τι βήματα θα λάβετε για να προχωρήσουμε προς μια νέα βιομηχανική πολιτική της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας. Ε, φυσικά θα είναι αδύνατο να καλύψετε όλες τις ερωτήσεις, ωστόσο νομίζω ότι είναι σημαντικό να ακούσει η Προεδρία τα θέματα που μας ενδιαφέρει να αντιμετωπίσει η Προεδρία. Στο σύντομο χρόνο που μας απομένει θα κάνετε ό,τι μπορείτε. Κυρία Υπουργέ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ αξιότιμοι ευρωβουλευτές για τις εξαιρετικές παρατηρήσεις και ερωτήσεις σας. Πολλές ερωτήσεις ακούστηκαν. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ομάδες. Ρωτήσατε σχετικά με την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη. Ε, όσον αφορά την ψηφιακή ε, οικονομία, σίγουρα θα συμπληρώσει τα λόγια μου η συνάδελφός μου, η κυρία Μαρίν. Πάντως, είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό για μας. Ε, θέλουμε να πετύχουμε νέα ανάπτυξη, κάτι που συνδέεται με την ερώτηση που τέθηκε. Επίσης σημαντικό είναι να έχουμε τεχνολογίες και τεχνικές ε, ώστε να έχουμε νέες μορφές ανάπτυξης. Όλα αυτά συνδέονται με το σχέδιο που έχουμε παρουσιάσει για μια ευρωπαϊκή βιώσιμη οικονομία. Τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά με το ορίζον Ευρώπη, τον προϋπολογισμό και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η κυρία να αναφέρθηκε στα θέματα αυτά κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Θα προσπαθήσουμε να οριστικοποιήσουμε αυτή τη δέσμη μέτρων. Κατά παράδοση, η Προεδρία δεν παρουσιάζει τις δικές της θέσεις. Ε, σημαντικό είναι να κλείσει το θέμα πάντως. Ε, όσον αφορά το ορίζον Ευρώπη, Σημαντικό είναι να έχουμε νέες τεχνολογίες και έρευνες ε, για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες ε, της ε, βιομηχανίας και να έχουμε ευημερία τους πολίτες μας. Χρειάζεται συνεργασία ανάμεσα στον πανεπιστημιακό χώρο και τις επιχειρήσεις. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε νέα ανάπτυξη χρησιμοποιώντας την έρευνα ανάπτυξη και καινοτομία ψηφιοποίηση, οικονομία των δεδομένων, η πτυχή της δεοντολογίας επίσης αναφέρθηκαν. Είναι σημαντικό σε όλες τις μελλοντικέ συζητήσεις να έχουμε ανθρωποκεντρική προσέγγιση, διότι εργαζόμαστε για το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Πιστεύω ότι η ψηφιοποίηση και οι νέες επιχειρήσεις ε, θα βοηθήσουν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας ε, να αναπτυχθούν. Τέθηκε μια γενική ερώτηση σχετικά με την εμπορική πολιτική. Είναι φυσικά απαραίτητο σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, να τονίσουμε την ανάγκη για μια παγκόσμια τάξη που να βασίζεται σε κανόνες. Έχουν δημιουργηθεί στρατηγικές ε, αλυσίδες αξίες για τις ευρωπαϊκές νεοφύης επιχειρήσεις. Ε, για παράδειγμα, ε, καθαρά αυτοματοποιημένα αυτοκίνητα, ανεξάρτητης οδήγησης και άλλα τέτοια θέματα, τα οποία θα σχολιάσει και η συνάδελφός μου. Όσον αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με το κλίμα το κλίμα είναι ένα πολύ ευρύ θέμα. Μπορώ όμως να πω ότι είναι ε, σημαντικό τα, ευρωπαϊκά, τα εθνικά στρατηγικά σχέδια να εκπονηθούν. Και με βάση αυτά να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένα μέτρα. Επίσης τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να πετύχουμε πρόοδο στις περιφέρειες. Τις νέες τεχνολογίες θα πρέπει να τις ε, αναπτύξουμε σε βιομηχανικό επίπεδο και είμαι βέβαιη ότι και άλλες περιφέρειες θα ενδιαφερθούν για αυτές αναφέρθηκε η δέσμη μέτρων για την καθαρή ενέργεια. Είναι σημαντικό να συνεχιστεί η συζήτηση το φθινόπωρο στο Συμβούλιο κατά την εξέταση των εθνικών σχεδίων για το κλίμα. Τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά με τα πυρηνικά απόβλητα και το σχετικό εναποθετήριο που έχει προβλεφθεί. Αναφέρθηκαν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις της Φιλανδίας, διότι είναι σημαντικό να έχουμε ασφαλή και υπεύθυνη διάθεση των αποβλήτων. Όσον αφορά το Εθνικό Σύστημα Ενέργειας ε, της Φιλανδίας, θα σας το παρουσιάσω σε διαφορετικό πλαίσιο, αλλά και αυτό είναι εθνικό θέμα. Εδώ εκπροσωπούμε το σύνολο του Συμβουλίου, δεν θέλουμε λοιπόν να μπούμε σε εθνικά ζητήματα. Σημαντικό είναι να παραμείνει υψηλό το επίπεδο φιλοδοξίας στην κλιματική πολιτική. Υπάρχουν όμως ε, κάποια ανησυχητικά φαινόμενα. Για παράδειγμα, αναφέρθηκε το πυρηνικό εργοστάσιο Αναστροβίτσε το... και είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει δράση και θα πρέπει να τηρούνται και οι διεθνείς συμφωνίες. Αναφέρθηκαν και οι ανησυχίες ε, που ε, σχετίζονται με τις ε, τουρκικές γεωτρήσεις στην ΑΟΖ της Κύπρου από τον κύριο Γεωργίου. Θα πρέπει να σκεφτούμε και το θέμα της ενεργειακής ένδυας. Αρκετοί ευρωβουλευτές αναφέρθηκαν στο θέμα αυτό. Έχουμε τις εκθέσεις των κρατών μελών για το, τα επίπεδα ενεργειακής ένδειας, όπως ανέφερε ο κ. Χέιζελ. Το ενεργειακό μείγμα είναι εθνικό θέμα. Έχουμε όμως ε, τους ε, κοινά συμπεφωνημένους στόχους για τη μείωση των εκπομπών. Πρέπει λοιπόν να μειωθεί η χρήση ορυκτών καυσίμων. Είναι σημαντικό να εφαρμοστούν μέσα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδυας από τα κράτη-μέλη. όσον αφορά την ψηφιακή επανάσταση και την κοινωνική αποδοχή κατά τη μετάβαση, είναι σημαντικό να εξετάσουμε τα διαφορετικά σενάρια. Ο κύριος Κέλλη ανέφερε στην παρέμβασή του το θέμα αυτό. και όσον αφορά τα εθνικά σχέδια για το κλίμα είναι μια ερώτηση στην οποία ήδη απάντησα στην προηγούμενη παρέμβασή μου. Θέλουμε να διασφαλίσουμε τα κράτη-μέλη να πετύχουν τους στόχους αυτούς και να τηρήσουν το πρόγραμμα. Είναι σημαντικό να υπάρχουν επαρκείς επενδύσεις ώστε να πραγματοποιηθεί επιτυχώς η μετάβαση. Δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, οπότε δεν μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις αυτή τη στιγμή. Τις κατέγραψα όλες όμως. Και θα τις λάβω υπόψη μου στη συνέχεια του κοινού μα ταξιδίου. Κάποιοι από εσά αναφέρθηκαν σε κοινοπραξίε στον χώρο της Έρευνα ανάπτυξη και κοινοτομία. Είναι σημαντικό να είναι ανοιχτές αυτές οι εταιρικέ σχέσεις, να διαφανείς, να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Να ευχαριστήσω την Πρόεδρο, να ευχαριστήσω και όλους σας για τις εξαιρετικές ερωτήσεις και παρατηρήσεις σας. Κλείνοντα να πω κάτι που αναφέρθηκε και σε πολλές άλλες παρεμβάσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συμμετοχή των πολιτών σε θέματα κλίματος και ενέργειας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να έρθω εδώ να σας μιλήσω. Ε, σημείωσα τις παρατηρήσεις σας και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια κατά τη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου, ώστε να έχουμε οικονομική ανάπτυξη, κοινωνικά και ε, οικολογικά δίκαιη και ε, έχουμε φιλόδοξους στόχους σε όλους τους τομείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις παρεμβάσεις, οι οποίες ήταν όλες ε, πολύ καλές. η συνεργασία και ο διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελπίζουμε ότι θα συνεχιστούν με καλό τρόπο. Ε, θα απαντήσουμε και γραπτό στις ερωτήσεις. Θα απαντήσω τώρα σε κάποιες ερωτήσεις που είναι τις αρμοδιότητές μου. Η κυρία Καρβάγιο ρώτησε για το 5G. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να σεβαστεί τις προθεσμίες που έχουν καθοριστεί για την ε, έναρξη λειτουργίας του 5G οι αρμοδιότητες ε, και οι γνώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο παγκοσμίω. Ρωτήσατε επίση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Υπήρξαν πολλέ ερωτήσει από αυτού. Τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ελήφθησαν μέτρα για να βελτιωθεί η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Για παράδειγμα, υπάρχει οδηγία και ο κανονισμό για τον τομέα αυτό και ε, η έχει μια νέα πιο ισχυρή εντολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ενισχύσει και να αναπτύξει την κυβερνοασφάλεια. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ε, την, ε, τον πανεπιστημιακό κλάδο, επιχειρήσεις. Προσπαθούμε να αντλήσουμε και διδάγματα από τα σφάλματά μας του παρελθόντος και ε, πιστεύω ότι η οδηγία για την ένισα είναι ένας ε, τρόπος να ενισχύσουμε όλα αυτά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να υπάρχουν περισσότερες διευκρινήσεις ε, τα κράτη-μέλη λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη όλα αυτά τα θέματα και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια καλή λύση. Είναι πολύ σημαντικό να δοθεί αρκετός χρόνος για συζήτηση ώστε το αποτέλεσμα να είναι όσο το δυνατόν καλύτερο. Όπως είπα, οι απειλές στον κυβερνοχώρο πρέπει να λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη και γίνονται πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή. Βεβαίως χρειαζόμαστε συνεχείς δράσεις, για παράδειγμα συνεργασία με αρχές επιβολής του νόμου, η οποία είναι πολύ έντονη από την αρχή της Προεδρίας μας. Προσπαθούμε να έχουμε συνεργασία με διάφορους ε, φορείς. Ε, ο κύριος Κρίστοφ ρώτησε για την ε, κλοπή προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει το GDPR που είναι το βασικό μέσο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Το Συμβούλιο παρακολουθεί ενεργά τις κλοπές στον κυβερνοχώρο. Μετά υπήρχε μια ερώτηση για την δίκαιη οικονομία στις πλατφόρμες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν σαφείς κανόνες, οι οποίοι θα είναι και δίκαιοι. Οι περισσότερες από αυτές τις ερωτήσεις βέβαια είναι χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Εργασίας. Ε, και στη συζήτηση για τα δεδομένα ελπίζω να μπορέσουμε να προωθήσουμε και τις αρχές ε, μιας δίκαιης οικονομίας δεδομένων. Ο κύριος Πούμπλιο ρώτησε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε η ψηφιακή ανταγωνιστικότητα να είναι εγγυημένη. Ε, πρέπει να δώσουμε έμφαση στο ίντερνετ των πραγμάτων, το 5G, την τεχνητή νοημοσύνη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε και νέα προγράμματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, στοιχείο εδώ. Οι τεχνολογίες αυτές πρέπει να χρησιμοποιηθούν, θα συζητηθούν αυτά ε, ιδιαίτερα ε, στο Συμβούλιο. Ε, υπήρχαν ερωτήσεις ε, ε, από την κυρία Λετάιο, τον κύριο ε, ε, Μάρκες για την ηλεκτρονική αναγνώριση ταυτότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε τη δήλωση. Για παράδειγμα, στο Ελσίνκι διοργανώνεται μια διάσκεψη τον Οκτώβριο για το θέμα αυτό. Η κυρία Λιτάιο Μάρκες ρώτησε επίσης ε, και για το πώς μπορούμε να περιλαμβάνουμε τους πάντες ε, ε, στην ψηφιοποίηση. Αυτό είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς θα συμμετέχουν οι πολίτες και νομίζω ότι η εκπαίδευση των πολιτών είναι η κατάλληλη λύση και φυσικά όχι λύση και φυσικά δεν είναι μόνο δική μου αρμοδιότητα, αλλά το πρόγραμμα της ψηφιακής Ευρώπης ε, προσπαθεί να τονίσει ε, και σε θέματα εκπαίδευσης ε, και το Συμβούλιο το έχει ψηλά στις προτεραιότητές του. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις του. Μπορεί να μην μπόρεσα να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Δεν είχα και επαρκή χρόνο στη διάθεσή μου, αλλά σίγουρα μπορούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας ε, και να είμαστε συνεχώς σε επαφή. Είμαι διατεθειμένη να επιστρέψω στην, στην Επιτροπή σας να συζητήσω αυτά τα θέματα και στο μέλλον βεβαίως και ελπίζουμε ότι θα είναι καρποφόρα συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και θα μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα τα οποία συζητήσαμε και σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τις δυο σας ε, για την παρουσία σας εδώ σήμερα και που μπήκατε στον κόπο να ακούσετε και να απαντήσετε σε ερωτήσεις μας. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για το ενδιαφέρον σε αυτή τη, για αυτή τη συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε στις 2.30 και κλεισμένο των θυρών ε, συνεδρίαση για το Καριλαίο. Καλή όρεξη.